κυρίες και κύριοι. Να αρχίσουμε. Ε, συντονιστής από το είναι εδώ. Θα μιλήσω ισπανικά. Πρώτο σημείο. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, σχόλια, τότε εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Δεν βλέπω καμία αντίρρηση εδώ, οπότε περνάμε στο δεύτερο σημείο που είναι τα πρακτικά τη Δευτέρα και 3η Οκτωβρίου 2019. Έχουν μοιραστεί τα πρακτικά σε όλα τα μέλη τη Επιτροπή μα. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, επίση θεωρούνται κεκριμένα. Δεν βλέπω αντιρρήσει, εγκρίνονται λοιπόν. Σημείο 3. Έχουμε εδώ πέρα διάφορε ανακοινώσει τη Προέδρου που ενημερώνει του Ευρωβουλευτέ για τα εξή. Πρώτον, ότι οι συντονιστέ ενέκριναν με γραπτή διαδικασία το πρόγραμμα το ερευνητικό το ετήσιο τη Επιτροπή μα. Το αποτέλεσμα τη γραπτή διαδικασία επίση όσον αφορά τα σημεία Β τη 4η και 5η Σεπτεμβρίου είναι τα εξή. Αναφορέ.

Οι αναφορές 0364 του 18, 0367, 0443, 0668, 0854, 0939, 984 και 1114 του 2018 παραμένουν ανοιχτές και θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη μιας επόμενης συνεδρίασης. Όσον αφορά την αναφορά 0420 2018 θα ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα στείλουμε επιστολές στην κεντρική κυβέρνηση της Ισπανίας αλλά και τις περιφερειακές. Επίσης, αναφορά 0649 2018 Πρόκειται για κοινή αντιμετώπιση με την αναφορά 0451-2008 και για την 08-27-18 θα ζητήσουμε περισσότερε πληροφορίε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 0902 θα συμπεριληφθεί σε μια επόμενη συνεδρίαση τη Επιτροπή μα και θα ενημερωθούν και οι αρμόδιες ισπανικέ αρχέ. Εντάξει. Ωραία. Ωραία. Τελειώσαμε το σημείο 3. Περνάμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Εδώ πέρα έχουμε δύο αναφορές. Την αναφορά 0676 κάθετος 2016 Πρόκειται για έναν πολίτη γερμανικής εθαγένειας σχετικά με την φερόμενη ω μονομερή και τη δημοκρατική νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μαζί με την αναφορά 0429 του 2017 του κυρίου Χάραλτ Μπόλσιγκερ Γερμανική ηθαγένεια σχετικά με τη συμμόρφωση τη Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προ το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε εδώ τους δύο αναφέροντε Σωστά, τον κύριο Σλομίσκι την, ε, και τον κύριο Χάραλτ Μπόλσιγκερ. Οπότε, εφόσον συμφωνείτε, θα δώσω πέντε λεπτά στον κάθε αναφέροντα. Συμφωνεί. Πρώτο κύριο κύριος Μπόλσιγκερ, παρακαλώ. Παρακαλώ κύριε Μπόλσιγκερ. Για πέντε λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, αξιότιμοι μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ, σε ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε την ε, αναφορά αυτή και δεχτήκατε να αναλάβετε παραπέρα βήματα. Ε, την βάλατε μαζί με την 0676 που στην ουσία δεν έχει καμία σχέση η μία με την άλλη. Θέλω να σας πω ότι εδώ δεν είμαστε για να ηθικολογήσουμε. Απλώς ζητούμε να σέβονται τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λοιπόν. Ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι εύκολο να το καταλάβει κανείς. Δεν βλέπω να λειτουργεί το σύστημα. Τέλος πάντων, ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι εύκολο να το καταλάβει κανεί, γιατί στα καθήκοντα και τι αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν, δεν περιλαμβάνεται λογοδοσία όσον αφορά την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι εδώ υπάρχει ένα κενό όσον αφορά την ηθική διάσταση που δεν περιλαμβάνεται στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία που έχουμε και έχουμε συλλέξει από διάφορες πηγές και κάθε φορά καταλήγουμε στα ίδια αποτελέσματα, ότι δηλαδή 20% των ε, λεγόμενων ε, αποδεκτών εμπορεύσιμων περιουσιακών ε, στοιχείων δεν περνάει από καμία τέτοια αξιολόγηση. Πρέπει να δείτε λιγάκι τον ε, όγκο εδώ πέρα, που είναι τεραστιο σχεδόν 14, ε, 14 ευρώ. Κάτι το οποίο πειράζει πάρα πολύ και την ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά και τους ευρωπαίους πολίτες. Έτσι λοιπόν τα κριτήρια επιλογής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις εγγυήσει που παίρνει έναντι πληρωμής και δανείων ή επενδύσεων ε, δεν περιλαμβάνουν τη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Δηλαδή είναι τυφλή όσον αφορά την ηθική διάσταση η χρηματοπιστωτική αγορά, όσον αφορά δηλαδή τις ευρωπαϊκές αξίες. Έτσι λοιπόν, τελικά αυτό το 20% που λέγαμε πριν παραβιάζει την ηθική. Και δεν υπάρχει και θέμα ανεξαρτησίας, γιατί αυτό είναι που λένε πολλοί ότι πρέπει να είναι ανεξάρτητη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όμω δεν υπάρχει καμία παραβίαση στην ανεξαρτησία τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αν αυτή συμμορφώνεται με τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Οπότε παρακαλώ, βοηθήστε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να συμμορφωθεί με τι ηθικέ αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δείτε την απάντηση τη ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει παρετέρω δράση. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί κανένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητο από τα θεμελιώδη δικαιώματα. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μην τι άλλο να δώσει κατευθυντήριες γραμμές για συμμόρφωση προς τις ε, θεμελιώδεις αρχές. Επίσης, εδώ γελάμε με αυτά τα κριτήρια ότι ας πούμε η αναφορά λέτε πρέπει να απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μα η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ζητάει από τις πολιτικές αρχές να ορίσουν, να συμφωνήσουν και να προωθήσουν ελάχιστες ηθικές προδιαγραφές. Για τη λογοδοσία επίσης της ε, ΕΚΤ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δίκιο μεν, αλλά θα έπρεπε να είναι σαφές ότι θα λογοδοτεί και για τα θεμελιώδη δικαιώματα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κάτι το οποίο δεν το έχει κάνει ποτέ να λογοδοτήσει σε σχέση με τη συμμόρφωσή τη στα θεμελιώδη δικαιώματα και εσείς μπορείτε να την αναγκάσετε να το κάνει να σας πει κατά πόσο συμμορφώνεται ή όχι στις δραστηριότητές της με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η συνθήκη της Λισαβόνας λέει ότι όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να εφαρμόζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα, άρα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η απάντηση τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δείχνει ότι περιμένει πολιτική δράση για να λυθεί αυτό το ζήτημα. Οπότε σα παρακαλώ, πραγματικά σα παρακαλώ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι θεματοφύλακα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Συνεπώ πρέπει να δράσει για την αναφορά αυτή. Και σα παρακαλώ να πείσετε την ΕΚΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διορθώσει αυτό το τεράστιο συστημικό λάθο που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα σε εσά είναι το μπαλάκι να σχεδιάσετε τα επόμενα βήματα εσείς πρέπει να αποφασίσετε τι θα κάνετε στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Σλομίσκι. Παρακαλώ. Εγώ αυτό που μπορώ να προσθέσω, μόνο στα γερμανικά, από τις 10 Δεκάτου 2019 έχετε μια, ένα γραπτό σημείωμα. Νομίζω ότι τα καλύπτει όλα. Η αναφορά είναι διεξοδικά τεκμηριωμένη. και δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά στο αιτιολογικό νομίζω ότι πρέπει απλώς να ληφθεί η σχετική ε, απόφαση. Βλέπουμε ότι η πολιτική των, της Ευρωπαϊκής Τράπεζα Τράπεζας απλώς... Ε, δεν αφήνει κανένα περιθώριο και νομίζω ότι στο γραπτό σημείωμα της 10 Οκτωβρίου 2019 λέγονται τα πάντα. Δεν χρειάζεται να το ε, επαναλάβω. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε τα γερμανικά. Ωραία, συνεχίζω στα γερμανικά. Το αντικείμενο της αναφοράς είναι οι αποφάσεις της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και είναι τιμωρητική η πολιτική επιτοκίων της ΕΚΤ, είναι αντιδημοκρατική και είναι μια πραγματική παραβίαση του βασικού δικαίου για το δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο, και δεν μπορεί να, συνδυαστεί με το σύνταγμα, να, είναι, να συνάδει το Σύνταγμα κανενός ε, κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ελέγχεται με ε, κατασταλτικό τρόπο χωρίς τα περιουσιακά στοιχεία των εθνικών κρατών να μπορούν να αξιοποιηθούν είναι πραγματική παραβίαση για τις νομισματικές αξίες που θέλουν τα κράτη-μέλη να προσπιστούν. Οι αποφάσεις λοιπόν της ΕΚΤ είναι κατά της οικονομικής και νομισματικής ε, λογικής και στην πράξη εφαρμόζεται μια πολιτική χωρίς ε, πραγματική ε, λειτουργία, χωρίς πραγματικό νόημα. Θα μπορούσε κανείς να αναφέρει μια παρήθμιση εδώ των αποφάσεων της ΕΚΤ που δημιουργούν προβλήματα στην πολιτική των κρατών μελών, αλλά η τιμωρητική πολιτική της ΕΚΤ δεν βασίζεται σε καμία πραγματική αρχή. Οι πολίτες στην Γερμανία αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα εξαιτία της προβληματικής αυτής πολιτικής της ΕΚΤ. Και ουσιαστικά καταπιέζονται τα βασικά τους, τα θεμελιώδη τους δικαιώματα ως προς την αξία των περιουσιακών τους στοιχείων. Αυτό είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να αναλάβουν δράση τα δημοκρατικά κράτη. Η τιμωρητική λοιπόν πολιτική επιτοκίων της ε, ΕΚΤΑ στην Ευρωζώνη είναι κάτι που θα έπρεπε να δουν τα κράτη-μέλη για να αναλυφθούν ευθύνες διότι η νομισματική και οικονομική πολιτική δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Η πολιτική και οι διαδικασίες που ε, προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέτρα δεν ε, ε, έχουν παρά μόνο αρνητικό και ακραίο αντίκτυπο γιατί καταστρέφονται οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων λόγω της πολιτικής της ΕΚΤ και ουσιαστικά δεν έχει καμία, κανένα πραγματικό στόχο η τιμωρητική αυτή πολιτική η, της ΕΚΤ θα έπρεπε να επιτραπεί στον γερμανικό λαό να διαθέσει ελεύθερα την, ε, να κανονίσει και να καταρτήσει ελεύθερα τη δική του πολιτική διότι έχουν ήδη ε, προκληθεί πολύ σημαντικές ζημιές, οικονομικές ζημιές. Ο αναφέρον λοιπόν ζητά να αναλυφθεί δράση κατά της ΕΚΤ διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εδώ ευθύνη. η κατάρτιση αυτής της πολιτικής από την Ευρωπαϊκή ε, Κεντρική Τράπεζα δεν περιορίζεται από κανέναν και θα πρέπει κάπως να αντιμετωπιστεί. Αναφέρονται αυτά διεξοδικά στο γραπτό σημείωμα της αναφοράς από τον αναφέροντα και ελπίζουμε να γίνουν αποδεκτά. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν συμφωνώ με την αναφορά αυτή, γιατί είναι μια εντελώ χωριστή αναφορά από την δικιά μου, λέει ο κύριο Μπόλσιγκερ. Πρόεδρο, αυτό θα το αποφασίσει ο πρόεδρο. Κύριε Σιμίσκι, βλέπετε έχει περάσει ο χρόνο σα. Είσαστε ήδη στα 6,5 λεπτά. Θα πρέπει να ολοκληρώσετε. Ωραία. Ε, εντάξει. Ολοκληρώσαμε και με αυτήν την αναφορά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα, παρακαλώ, ο κύριος Ματέος Σάλτο. Χαίρετε. Θα μιλήσω αγγλικά εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Ευχαριστώ και τους δύο αναφέροντες. Οι δύο αυτές αναφορές πράγματι είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Θα ξεκινήσω με τη δεύτερη αναφορά ίσως, την 0676. Ε, σε σχέση τώρα με την προηγούμενη ακρόση, ποια είναι η διαφορά. Είναι η επιστολή του αναφερόμενου του Οκτωβρίου φέτος. Τη συνόψεις ουσιαστικά. Εμείς πιστεύουμε ότι το συμπέρασμά μας δεν αλλάζει. Δηλαδή πιστεύουμε πράγματι ότι πρέπει να απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το, ο, το μόνο που θέλουμε να τονίσουμε εδώ είναι ότι στο μεταξύ υπήρξε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που είπε ότι το πρόγραμμα αγοράς δημοσίων ομολόγων ευθυγραμμίζεται με τις συνθήκες. Αυτό είναι το μόνο νέο στοιχείο που έχουμε. Κατά τα άλλα δεν αλλάζει τίποτα, οπότε δεν αλλάζει ούτε η τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έρχομαι τώρα στην άλλη αναφορά, την 0429 του 2017. Και πάλι ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή της. Τώρα, ενώ συμφωνούμε με ότι όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεσμεύονται από τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, όμως πιστεύουμε ότι ως αρχή που απορρέει από τον νόμο, η εφαρμογή της χάρτας αυτής δεν τροποποιεί τις αρμοδιότητες έτσι όπως αυτές διατυπώνονται στη συνθήκη. Η αναφορά αυτή βέβαια δεν είναι για την Κομισιόν, για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οπότε εμεί απλώς επιβεβαιώνουμε την αρχή αυτή. Διότι η πολιτική όσον αφορά τις ε, διάφορες ε, πολιτικές ε, ε, προγράμματα κτλ. Είναι πράγματα τα οποία διέπονται από την συνθήκη. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Οι συντονιστές τώρα, παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Κίλτον Ντάρλινγκ. Να συμφωνήσω με τον αναφέροντα τον κύριο Μπόλσιγκερ. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικές οι αναφορές μεταξύ τους. Και βρίσκονται μένει υπό το ίδιο σημείο στην ενίσχυση διαταξή, αλλά καλό θα είναι να πούμε κάτι διαφορετικό για την καθεμιά τους. Ε, προφανώς στο Ευρωκοινοβούλιο γίνεται έντονη συζήτηση για την ε, πολιτική, την νομισματική πολιτική της ΕΚΤ. Η συζήτηση αυτή λαμβάνει κυρίως χώρα στην Επιτροπή ΕΚΟΝ Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων και σε συνεννόηση με την την ίδια, με πολύ συστηματικές ανταλλαγές. Οπότε, εάν ακόμη δεν έχουμε παραπέμψει, αναπέμψει μάλλον τις αναφορές στην Επιτροπή ΕΚΟΝ, καλό θα ήταν να το κάνουμε, για να τις ε, χρησιμοποιήσουμε στις επόμενες συζητήσεις μας. Η θέση μου τώρα Νομίζω το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της συμμόρφωσης με αυτά είναι ενδιαφέρον. Αυτό αυτό. Δηλαδή να δούμε σε τι βαθμό η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων καλύπτει όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένε της ΕΚΤ, και ε, επειδή συζητάμε σε διαφορετικέ επιτροπέ για την Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα, α πούμε, και τα κριτήρια που χρησιμοποιεί, η συζήτηση που γίνεται είναι συνήθω έντονη για το πώ ε, είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει συμμόρφωση με τι ευρωπαϊκέ αξίε στα διάφορα θεσμικά όργανα, στα διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ούτω καθεξής. Οπότε νομίζω ότι καλό θα ήταν και από τη δική μας την πλευρά να στείλουμε την αναφορά στον νέο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής, στη νέα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η αναφορά για τα θεμελή δικαιώματα να παραμείνει ανοιχτή διότι είναι μέρος μιας συζήτησης που θα συνεχιστεί και στο μέλλον στην Επιτροπή ΕΚΟΝ και θα μπορούσαμε λίγο να δώσουμε μια συνέχεια στα συγκεκριμένη αναφορά στις συζητήσει μας εδώ στο Κοινοβούλιο και στην συγκεκριμένη Επιτροπή. Από την απάντηση της Επιτροπής τώρα καταλαβαίνω ότι το βασικό σημείο που θέτει η πρώτη αναφορά, η 676, για την έλλειψη συνταγματικού ε, χαρακτήρα συνταγματικών αρχών στον τρόπο που καταρτίζει τις πολιτικές της η ΕΚΤ έχει επιληθεί και απαντηθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εάν είναι λοιπόν έτσι, ε, φαίνεται ότι έχει κλείσει το βασικό σημείο που έχει η αναφορά, οπότε θα πρότεινα να κλείσει η αναφορά και θα έλεγα να αντιμετωπίσουμε τις δύο αναφορές με διαφορετικό τρόπο όπως τους αρμόζει. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ. Και εγώ νομίζω ότι πρέπει να τις δούμε διαφορετικά τις δύο αναφορές. Εάν κατάλαβα καλά την συνάδελφο, ποια λέτε να μείνει κλειστή και ποια, ποια λέτε να κλείσουμε και ποια να μείνει ανοιχτή. Την πρώτη να κλείσουμε και την άλλη να την αφήσουμε ανοιχτή ή αντίστροφα. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση θα τα δούμε ξεχωριστά, διότι αφορούν διαφορετικά θέματα για την αναφορά του κυρίου Μπόλσιγκερ. Πολιτικά το θέμα είναι και ευαίσθητο και πολύ ενδιαφέρον και πραγματικά θα πρέπει να δούμε την ΕΚΤ και σε αυτή τη διάσταση. Πολλές φορές Θα πρέπει να μπορεί να αποδειχθούν κάποια πράγματα στην οικονομική και νομισματική πολιτική και τις αποφάσεις τους. Οπότε νομίζω ότι η συζήτηση αυτή και ευαισθητή είναι και μπορεί συνέχεια να έχει. Τώρα, κατά πόσο ανάπτυξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων το θέμα αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε και όντω θα πρέπει να αναλάβει η υπεύθυνη επιτροπή. Θα πρέπει να λάβουν γνώση επίση και η υπεύθυνη τη ΕΚΤ. Τώρα για την άλλη αναφορά. για την 161 και εκεί τα θέματα είναι σημαντικά και ευαίσθητα. Και εκεί υπάρχουν πολιτικές προεκτάσεις. Και δημοσίωση ΕΚΤ, κατά την άποψή μου, έχει αναγνωρίσει εν μέρη τις ευθύνες της εδώ και το θέμα θα μπορούσε να κλείσει. διότι το ένα θέμα άπτεται της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, το άλλο όμως ε, έχει απαντηθεί νομικός, οπότε θα μπορούσε και να κλείσει. Ευχαριστούμε κυρία Μίλλερ. Ναι. Και εγώ θα ήθελα να μιλήσω εξ ονόματος της συντονίστριας που δεν μπορεί σήμερα να είναι εδώ και να συμφωνήσω με τον κύριο Γιάρ Ίσως ο συνάδελφος από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες κάτι να μην ε, κατάλαβε σωστά. Εγώ Εγώ κατάλαβα ότι η Επιτροπή 04 ε, 2 θα πρέπει να ε, λάβει συνέχεια γιατί έχει να κάνει με θεμελιώδη δικαιώματα. Είναι σημαντικό ε, θέμα που θα μπορούσε να μας απασχολήσει. Για την δεύτερη δεν μπορώ να το φανταστώ γιατί ξέρω ότι στην Γερμανία είναι πολλοί οι απλοί πολίτες που είναι εξοργισμένοι για τις οικονομίες τους και τον τρόπο που έχουν αποταμιεύσει και για το πώς τις έχουν μεταχειριστεί με τις ε, πολιτικές τους από την ΕΚΤΑ. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και νομίζω ότι έχει κλείσει, θα μπορούσε να κλείσει αναφορά αυτή. Ευχαριστούμε. Οι αναφέροντες. Δύο λεπτά, λεπτά καθένα, παρακαλώ. Ο κύριο Βόλιγκερ πρώτα. Δεν κατάλαβα ποια είναι η ερώτηση. Έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή σας ε, για να κλείσετε σχετικά με την ε, αναφορά. Δεν θέλω να την κλείσω, την αναφορά. Δεν καταλάβατε τι εννοώ. Εννοώ να πείτε κάποια σχόλια συμπερασματικά για να κλείσουμε το σημείο της ημέρης διάταξης. Όχι για να κλείσετε τελείως την αναφορά. Εσείς, ε, κύριε Φεράρα, είμαι πολύ ικανοποιημένο που τα είπατε αυτά, γιατί εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε θεματοφύλακες των δικαιωμάτων αυτών και αναρωτιέμαι ποια θα είναι τα επόμενα βήματα που θα κάνετε και τι θα σας απαντήσει η Κριστιαν Λαγκάρτ ή τι μπορεί να κάνει σε αυτή την περίπτωση. Αν μπορώ λοιπόν με οποιοδήποτε τρόπο να σας βοηθήσω, σας παρακαλώ πείτε το μου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σλομίνσκι για δύο λεπτά. Äh, Τι να προσθέσω τώρα. για όσα προκύπτουν από τη διαδικασία της αναφοράς είναι σαφές ότι η ΕΚΤ δεν είναι ανεξάρτητη από την Ένωση στο πώς λαμβάνονται τις αποφάσεις. Είναι όλα αντικανονικά και ε, προσβάλλονται τα δικαιώματα των πολιτών γιατί είναι τιμωρητική η πολιτική επιτοκίων στο νομισματικό χώρο της Ευρωζώνης. Οπότε θα έπρεπε, μάλλον αυτό που συμβαίνει επίσης λόγω της ε, πολιτικής των επιτοκίων της ε, ΕΚΤ, θα έπρεπε να υπάρξει και αποζημίωση για αυτήν την ε, πολιτική δεν θα πρέπει να παραμείνει ε, στη διάθεση της ΕΚΤ αυτή η ελευθερία να καταρτίζει την πολιτική όσο έχει και να επιφέρει ζημιές και είναι θέμα ε, αρχής. Η τιμωρητική λοιπόν ε, πολιτική επιτοκίων είναι πραγματική παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και είναι και το πραγματικό αντικείμενο της αναφοράς, η προσβολή αυτών των βασικών αξιών. Δεν ξέρω αν κάτι μου διέφυγε εδώ, θα πρέπει να τα ψάξω λιγάκι μες στο κείμενο. Είναι σωστά αυτά μεταξύ άλλων στην απάντηση της ΕΚΤ λέγεται ότι οι βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποτίθεται ότι κατοπτρίζονται από, στην πολιτική της ΕΚΤ, όμως οι παραβιάσεις είναι πραγματικά καθημερινές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα αξιόγραφα που εκδίδει επηρεάζει ουσιαστικά επηρεάζει την πολιτική της. Με συγχωρείτε κύριε Σλοβίνσκι, αλλά πρέπει να ολοκληρώσετε. Τι λέτε? Πρέπει να ολοκληρώσετε. Μπορείτε να το επαναλάβετε. Τι, τι είπατε? Α, καλά. Δέκα δευτερόλεπτα. Για να αλλάξει λοιπόν αυτή η κατάσταση θα πρέπει να γίνει παραδεκτή η αναφορά και να ληφθεί δράση με τις ανάλογες πολιτικές διαδικασίες του Ευρωκοινοβούλιο, διότι η ΕΚΤ και όλοι οι υπεύθυνοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να επιτρέψουν ε, τις, τις ε, εμπορικές τράπεζες να ακολουθήσουν τις υποχρεώσεις. Τελεία. Αυτό είναι το αντικείμενο της αναφοράς. Τέλος. Ακούσαμε λοιπόν τους δύο αναφερόμενους και ακούσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως επίσης και τους συντονιστές, βουλευτές, από τις διάφορες ε, πολιτικές ομάδες. Προτείνουμε λοιπόν η αναφορά αυτή την οποία έχει υποβάλει ο κύριος Σλοβίνσκι, η 0 δηλαδή 676 του 2016, Προτείνουμε λοιπόν ε, η αναφορά αυτά που έχει αρμοδιότητα αποκλειστική Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μια και είναι ένα εξάρτητο όργανο σύμφωνα με τη συνθήκη, προτείνουμε λοιπόν στον αναφερόμενο να απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στην Τράπεζα της Γερμανίας, την Bundestag, και αν συμφωνούν οι συντονιστές, κλείνουμε αυτή την αναφορά. Τώρα για την δεύτερη η οποία είναι η 0429 του 2017 του κυρίου Χάραλ Μπόλσιγκερ. Εδώ θα την αφήσουμε ανοιχτή. Ακούσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους συντονιστές και λαμβάνοντας υπόψη πως έχουμε καινούρια ε, διοικήτρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα την αφήσουμε ανοιχτή. Θα στείλουμε μία επιστολή στην Επιτροπή ε, ΕΚΟΝ, το έχουμε ήδη κάνει, και μας απάντησε πως έχει ήδη ζητήσει να αυξηθεί η διαφάνεια στα θέματα οικονομικής και νομισματικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και γίνεται ένας διάλογος ε, ε, που συνεχίζεται μεταξύ Προέδρου της ΕΚΤ και Επιτροπής ΕΚΟΝ. Γι' αυτό θα στείλουμε μια επιστολή στην ΕΚΤ με την ε, αναφορά του αναφερόμενου και αυτό θα λάβει και πάλι υπόψη την νέα Πρόεδρο της ΕΚΤ. Αυτά αποφασίσαμε για το συγκεκριμένο σημείο. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αναφερόμενους οι οποίοι παραβρέθηκαν τη σημερινή συνάντηση. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 5. Είναι μια αναφορά που έχει υποβάλει ο Αλμπέρτο Αράντ Σανταντέρ, υπήκος Ισπανίας, είναι η 0161 του 2017 για τις τραπεζικές πρακτικές της ΕΚΤ. Είναι εδώ ο κύριος Αράνς, οπότε για 5 λεπτά έχει το λόγο. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ ε, και χαίρομαι που δίνετε φωνή στους πολίτες. Την πρώτη φορά που ήρθαμε στην Επιτροπή Αναφορών μας είπαν πως η πρότασή μας ε, δεν θα... Ε, συζητηθεί. Αυτή τη φορά ήρθαμε πιο πολύ με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και έχουμε αυτή τη στιγμή εκπροσώπους από τη Βαλένσια, ε, από την Οριχουέλα και από την ευρύτερη περιοχή ε, για τις οικογένειες που έχουν επηρεαστεί από αυτή την σε εισαγωγικά κρίση, που είναι οι πραγματικοί πατριώτες στη χώρα μου. Για χρόνια προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι ακριβώς κρύβεται πίσω από αυτή την ε, πρακτική ε, και το σκοταδισμό που περιβάλλει αυτή την πολιτική. Γνωρίζουμε λοιπόν τι έχει συμβεί, γιατί έχουμε μιλήσει με πάρα πολλές ομάδες σας παρακαλώ πολύ να μιλάτε πιο αργά για να μπορούν να σας μεταφράσουν. Ναι, συγγνώμη, λυπάμαι. Κάναμε λοιπόν μια μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης και στα δικαστήρια και στην κοινή γνώμη. Στείλαμε αναφορές ε, και σε πολίτες και σε ενώσεις πολιτών ε, και στους δήμους εκατοντάδες σε όλη την Ευρώπη και μου κάνει εντύπωση γιατί είναι τα πολιτικά κόμματα τα οποία ε, αφήνουν χωρίς φωνή ε, ανθρώπους που θα μπορούσαν να παραστούν στο ε, δικαστήριο και να υπερασπιστούν αυτούς οι οποίοι χρωστάνε. Είναι μέθοδοι που δεν είναι... Είναι πρακτικές, με συγχωρείτε, οι οποίες δεν είναι θεμητές. Πάρα πολλές φωνές ακούστηκαν στο Αλικάντη, στη Σεβίλη, στη Ματρίτη, στη Βαρκελόνη ε, καταθέσαμε μία αναφορά με πολλές τροπολογίες από όλες τις πολιτικές ομάδες στη δική μας Βουλή. Αλλά δυστυχώς, παρόλα αυτά, δεν είχαμε τα αποτελέσματα που απαιτεί από μας η κοινωνία. Ζητήθηκε λοιπόν να αλλάξουμε τους κανονισμούς έτσι ώστε το δικό μας αίτημα να είναι πιο αποτελεσματικό ε, ενώπιον των δικαστηρίων. Στην ε, Εξτρεμαδούρα υποχρεώνονται οι τράπεζες να μας δώσουν τις πληροφορίες που ε, απαιτούμε. Μετά το ίδιο συνέβη στην και μετά στην ε, περιφέρεια της Βαλένσια. Είναι λοιπόν ε, ένα ε, καθεστώς για τον καταναλωτή που καλύπτει την αυτόνομη περιφέρεια της Βαλένσια και δίνεται ενημέρωση για τις υποθήκες χωρίς να τίθεται θέμα τραπεζικού απορρίτου. Εμείς αυτό το έχουμε ζητήσει ε, από όλες ε, από όλε τι τράπεζε, γιατί θέλουμε ο καταναλωτής να μπορεί να ενημερωθεί για όλα τα στοιχεία που καλύπτουν την υποθήκη του. Το ζητήσαμε από το 2016 και έχουμε το σχετικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε και από το, Δεκέμβριο, ε, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2 Δεκεμβρίου του 2017 και ευτυχώς, επειδή έχουμε ε, δικηγόρους που μας ε, εκπροσωπούν, καταφέραμε στη δική μας αυτόνομη περιφέρεια η εισαγγελία να συνταχθεί μαζί μας. Η Ένωση Καταναλωτών ε, μιλά για 15.000 τέτοιου είδους αιτήματα που έγιναν για προστασία πρώτης στέγης για σπίτια τα οποία κινδύνευαν και τα περισσότερα από αυτά που τα οποία έτυχαν δικαστικής προστασίας βρίσκονται στην περιφέρεια της Βαλένσιας. Ε, υπάρχουν πάρα πολλές προσπάθειες που γίνονται κρυφά από τους καταναλωτές με αποτέλεσμα ε, να ε, μην γίνεται σεβαστό το δικαίωμα ε, κυδαιμονίας που υπάρχει ε, στα δικαστήρια και τι συμβαίνει στα δάνεια που ε, ή που ε, δεν αποπληρώνονται, χάνει τον τίτλο και την κατοχή του δανείου η τράπεζα και την αναλαμβάνει κάποιο ανεξάρτητο ταμείο. Δηλαδή, δεν είναι πιστωτής πια η τράπεζα, αλλά είναι μόνο διαχειριστής και δεν μπορεί να απαιτήσει ε, στο δικό της όνομα η τράπεζα να πληρωθούν οι δόσεις που δεν έχουν πληρωθεί. Το Υπουργείο Οικονομικών το Σεπτέμβριο είπε πως σε τέτοιου είδους ε, δίκη ε, θα παρέμβει για πρώτη φορά και αυτό αποτέλεσε για μας ένα κομβικό σημείο. Το γεγονός δηλαδή ότι η Οικονομική Εισαγγελία αποφάσισε να ε, παρέμβει σε τέτοια περίπτωση υποθήκης που δεν πληρώνεται. Ξέρετε ότι πάρα πολλοί κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει πια τις δόσεις. Και θέλουμε να υπενθυμίσουμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πως το βασικό του καθήκον είναι να υπαγρυπνά για την οικονομική σταθερότητα και για τα πιστοτικά ειδήματα, τα οποία θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να διατηρείται η σταθερότητα ακριβώς του τραπεζικού συστήματος. Αν λοιπόν αυτές οι, αυτά τα αιτήματα που έχουμε καταθέσει ε, στην ε, Ισπανία ε, δικαιωθούν, ε, μπορεί να ακολουθήσουν χιλιάδες αγωγές οι οποίες θα πλήξουν για μια φορά ακόμα την αξιοπιστία του τραπεζικού μας συστήματος. Έχετε λοιπόν μια χρυσή ευκαιρία να απεγκλωβιστείτε από αυτή την κατάσταση και να φανείτε πως εσείς προστατεύετε όντως τη σταθερότητα του συστήματος. Ευχαριστούμε πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κ. Λαμάρκα παρακαλώ. Υπάρχει κι άλλος αναφέρον εδώ. Υπάρχει... Άλλα πέντε λεφτά μπορείτε να έχετε, γιατί υπάρχει και άλλη αναφορά. Αν θέλετε μπορείτε να μοιραστείτε το χρόνο. Αλλά έτσι κι αλλιώς και μετά στα συμπεράσματα ίσως μπορεί ο αναφέρον πάρει το λόγο και πάλι. Τι λέτε, τι θέλετε. Συμφωνείτε, ωραία. Τότε θα δώσουμε τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στον κύριο Μάρκο Λαμάρκα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω αγγλικά, αν δεν σας πειράζει. Άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την παρουσίαση και την ευχαριστώ πολύ την αναφέρουσα για την παρουσίαση αυτή. Πράγματι, το θέμα δεν είναι θέμα ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Βλέπετε, είναι θέμα αστικού δικαίου, καθαρά. Και αυτό σημαίνει ότι οι εθνικές αρχές είναι εκείνες οι οποίες νομοθετούν για τέτοιου είδους ζητήματα. Και απόδειξη αυτού είναι ότι η Εθνική Αρχή, η Τράπεζα της Ισπανίας και το Αρμόδιο Υπουργείο λένε ότι πηγαίνει η υποθήκη με το χρέος στα funds. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν καλύπτει αυτή την πτυχή. Και πράγματι πρέπει να σας πω ότι αν με τη μεταφορά του χρέους μεταφέρονται και προσωπικά δεδομένα, τότε σύμφωνα με τον κανονισμό για την προστασία ε, προσωπικών δεδομένων θα έπρεπε οι ενδιαφερόμενοι να είχαν ενημερωθεί. Τα δεδομένα όμως δεν μεταφέρονται για την προστασία ακριβώς των καταναλωτών. Ε, το μόνο που θα μπορούσα να πω νομοθετικά είναι ότι υπάρχει ενεξέλιξη η αναθεώρηση της οδηγίας για τα ανεπόθηκα δάνεια. Και έτσι μπορεί να αλλάξει κάτι. Αλλά προς το παρόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει τίποτα για αυτό το θέμα προστασίας των καταναλωτών. Ευχαριστούμε πολύ. Οι πολιτικές ομάδες τώρα. Πίτερ Γιάρ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αξιοσημείωτη. Ακούμε ότι θέλουμε την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου, πολύ καλά διατυπωμένο αυτό, αλλά ότι το θέμα της αναφοράς είναι θέμα του εθνικού δικαίου και ότι τα ενυπόθηκα δάνεια έχουν να κάνει με τη χώρα μέλος. Όμως η τελευταία φράση δείχνει ότι αν εγώ έχω μια υποθήκη από μια τράπεζα δεν θα πρέπει να ξέρω μετά με ποιον διαπραγματεύομαι, ποιος είναι ε, από την άλλη πλευρά για να διαπραγματευτώ. Οπότε πολύ ενδιαφέρουσα η τελευταία πρόταση που ακούσαμε. Και όντως στην πολιτική η πραγματικότητα έχει μεγάλη σημασία. Τα δεδομένα όντως πρέπει να είναι ανώνυμα, αυτό λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά θα πρέπει να ξέρω με ποιον συναλλάσσομαι. Και αυτές οι υποθήκες που έχουν τιτλοποιηθεί και περνάνε από τον ένα στον άλλον έχουν σαν αποτέλεσμα τελικά ο καταναλωτής να μην ξέρει με ποιον έχει να κάνει. Ήταν ενδιαφέρον που άκουσα την Επιτροπή να λέει ότι θα πρέπει να το δούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να δούμε τι γίνεται με τις υποθήκες και την οδηγία αυτή για τις υποθήκες. Θα έλεγα να το πάμε το θέμα στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Κάτι θα έπρεπε να γίνει εδώ. Οπότε, θα πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει τον κανονισμό για τις υποθήκες. Οπότε, τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον, έτσι όπως έχει σήμερα η κατάσταση. Προφανώς δεν μπορούμε να πούμε στον αναφέροντα «Α, τελείωσε, εμεί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, είναι η χώρα μέλος, ακόμα και αν ξέρουμε ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο καλή». Στο κάτω-κάτω και άλλοι έχουν το ίδιο πρόβλημα. Οποιοδήποτε που έχει μια υποθήκη, ξαφνικά η άλλη πλευρά αλλάζει και δεν ξέρουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Λοιπόν, με τη σημερινή κατάσταση, ναι, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τον αναφέροντα, αλλά μπορούμε να ζητήσουμε από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή να κοιτάξει το θέμα, να δει μήπω κάτι πρέπει να αλλάξει. Και να έχουμε ένα διαφορετικό τελικά πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω αυτό πρέπει να είναι το συμπέρασμα, ότι από τη μια λέμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω από τη, για την αναφορά και μπορεί και να κλείσει, αλλά να πάει το θέμα στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί δεν μπορεί να κρύβονται πίσω από τον κανονισμό για την προστασία των ε, δεδομένων ε, διάφορα funds και να μην ξέρουμε ποιοι είναι. Σήμερα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αλλά μπορούμε να κάνουμε μια προσπάθεια να αλλάξουμε τα πράγματα για το μέλλον. Και αν κατάλαβα καλά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης, αν μη τι άλλο, το σκέφτεται ότι ίσως θα μπορούσε να αλλάξει η κατάσταση. Αυτό να είναι το σημείο κίνηση Η κυρία και τον Darling. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα σχολιάσω τα όσα είπε ο Πίτερ και θα διαφωνήσω ελαφρώς με τη δική του σύσταση. Πραγματικά με παραξένεψε η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουν περάσει 12 χρόνια από το οικονομικό κράς που είχε να κάνει με την τίτλοποίηση υποθηκών και η απάντηση πως είναι αρμοδιότητα εθνική και ενδεχομένως ότι θα το δούμε όταν αναθεωρηθούν οι κανόνες περί προστασίας καταναλωτών με την υπόθηκα δάνεια μου είναι αδιανόητο ότι η κατάσταση δεν έχει ε, τοποθετηθεί στον πυρήνα των αναθεωρήσεων που θα κάνουμε στην Ευρώπη για τους ε, σχετικούς κανονισμούς δεδομένων των κινδύνων που κρύβουν αυτά τα επικίνδυνα ε, προϊόντα και η τιτλοποίηση των υποθηκών έχει πλήξει χιλιάδες κόσμου στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ η προστασία του καταναλωτή και η νομοθεσία για τα ενυπόθηκα δάνεια είναι ένα θέμα που μας αφορά. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές αναφορές από τη Βουλγαρία για την προστασία των καταναλωτών με αυτή τη νομοθεσία. Ξέρουμε πως σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχουν τέτοια προβλήματα και γίνεται μια συνεχής αναθεώρηση της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας Οπότε θα ήταν πολύ σημαντικό εμείς ως Επιτροπή να δούμε πώς μπορούμε αυτές τις αναφορές να τις προωθήσουμε, γιατί τονίζουν διαφορετικά θέματα στα διαφορετικά κράτη-μέλη, αλλά ανήκουν στην ευρύτερη ε, διάσταση του προβλήματος, έτσι ώστε να το κάνουμε με έναν τρόπο που να εξασφαλίσουμε πως η δική μας νομοθεσία θα ανταποκρίνεται στις ανησυχίες των πολιτών. Είμαι πέντε χρόνια στην Επιτροπή Αναφορών και είχαμε προφορικές ερωτήσεις για την κατάσταση στην Ισπανία, στην Ολομέλεια, ε, ψήφισμα για τα στεγαστικά στην Ισπανία. Ήταν πολύ ωραία λοιπόν που ακούσαμε από τους αναφερόμενους το τι συμβαίνει στην Ισπανία με τις τοπικές δράσεις που έχουν λάβει. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω γιατί είναι ωραία να ακούμε και καλά νέα στην Επιτροπή μας. Αυτό πρέπει να το πούμε. Το ζήτημα αυτό δεν έχει κλείσει. Πιστεύω η αναφορά πρέπει να μείνει ανοιχτή και ίσως να σκεφτούμε εμείς αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη δική μας, το δικό μας δυναμικό για να ζητήσουμε μία αναφορά ή μία μελέτη για το θέμα αυτό Πολλές σχετικές αναφορές έχουμε ακούσει από κράτη-μέλη και να δούμε πώς μπορεί σε αυτές οι ανησυχίες που εκφράζονται να χρησιμοποιηθούν για να βελτιωθεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό για μια επόμενη συνάντηση των συντονιστών. Ευχαριστώ πολύ. Παρόλο, λοιπόν, αφού δεν υπάρχουν άλλες πολιτικές ομάδες που να θέλουν να πάρουν το λόγο, θα ζητήσω από τον κύριο Ράντς σε δύο λεπτά να αναφερθεί. Με συγχωρείτε ε, που παραμένω στο θέμα Σα ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο και θέλω να υπενθυμίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πω αυτά τα φάνη που τυκλοποιούνται τα έχει αποκτήσει η αναφορά μα βασίζεται στο γεγονός πως αυτά τα funds που τιτλοποιούνται τα έχει αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και γι' αυτό εμείς αναφερθήκαμε σε εσά. Όλοι γνωρίζουμε πως ε, το ξέπλυμα είναι ε, έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΚΤ προσπαθεί να συνεργαστεί με τις κρατικές τράπεζες για να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Γίνεται από μεγάλες επιχειρήσεις και κάνουν προσπάθειες για να συνεργαστούν με τις εθνικές αρχές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην επιστολή που μας έστειλε ο κύριος Νομπλέτ 23 Ιανουαρίου του 2018 είπε πως ο κανονισμός ε, MUS βασίζεται στους προηγούμενους ε, κανονισμούς τον 1024 από το 2013 όπου ζητά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να δώσει μια συγκεκριμένη πολιτική ε, πολιτική απόκριση στην προληπτική εποπτεία των χρηματοπιστικών ε, ιδρυμάτων και θα πρέπει όπου ενδεδειγμένο να συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες ώστε να υπάρχει το κατάλληλο επίπεδο προστασίας του καταναλωτή και η καταπολέμηση του ξεπλήματος. Η... Τα δικαστήρια στην Ισπανία έχουν ε, εκδώσει αποφάσεις όπου ε, τα χρηματοστοπιτατικά αυτά φαντ ε, μοιάζουν να διαχειρίζονται και να έχουν στην κατοχή τους αυτά τα ενυπόθηκα δάνεια. Και σε πολλές περιπτώσεις αυτό το έχει χαρακτηρίσει ως ποινικό αδίκημα. Ε, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε πάρα πολλές παραβιάσεις, αλλά για να το αποδείξουμε πως δεν είναι κάτοχος του τίτλου έπρεπε να βρούμε ανάμεσα σε αυτά τα φαντ. Κύριε Ράντς, πρέπει να μιλάτε λίγο πιο σιγά για τους διερμηνείς. Έτσι κι αλλιώς έχει λήξει ο χρόνος σας, θα σας δώσω 20 δευτερόλεπτα, αλλά σας παρακαλώ πολύ πιο σιγά. Οι δύο επιστολές λοιπόν μας έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάνε για το τραπεζικό απόρριτο και το γεγονός της σεβασμού της ιδιωτικότητας, ε, της αλληλογραφίας ε, άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λάβουμε κανένα στοιχείο για κανέναν επενδυτή, για κανένα φαντ, για κανέναν οτιδήποτε. Εμείς όμως ε, ε, ζητάμε κάτι διαφορετικό και γι' αυτό που μου κάνει εντύπωση που επικαλείστε την ανωνυμία. Ζητάμε τα δικά μας στοιχεία και οι τράπεζες τα έχουν γιατί έχουμε συμπληρώσει τα σχετικά στοιχεία σε αιτήσει μας. Θέλουμε λοιπόν για κάθε ένα ε, υπόθηκο δάνειο να μας πει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα τι έχει συμβεί με την τιτλοποίησή του. Στο κεφάλαιο 3, όπου μιλάμε για τα μητρώα ε, ε και για το μητρό των φανς που μπορούν να αναλάβουν αυτά τα καθήκοντα, μιλάνε και για κοινοποιήσεις σχετικά με το θέμα αυτό ε, και με όλα τα στοιχεία που είχαμε ε, στην έκθεση του Συμβουλίου Παριθμών 78 με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του ποινικού και διοικητικού δικαίου για άτομα τα οποία δεν είναι αρμόδιες αρχές και που λαμβάνουν απόρριτες πληροφορίες θα πρέπει αυτό να λαμβάνει υπόψη τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους χωρίς αυτό να παρακολεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για όλα τα θεσμικά όργανα τα οποία έχουν ως καθήκον να προστατεύσουν ε, ε, την ε, σχετική ε, νομοθεσία να λαμβάνουν τα στοιχεία αυτά και αυτό θα μπορούσε να είναι θεσμικά όργανα όπως για παράδειγμα το Ανώτατο Συμβούλιο για τα Τραπεζικά Θέματα ε, το οποίο έχει και τις αρμοδιότητες του Εθνικού Μητρώου και στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι όλοι αυτοί οι κατανοητές. Κύριε Αράνς. Κοιτάξτε, <clears throat> έχει περάσει ο χρόνος. <clears throat> Πέντε δευτερόλεπτα ακόμα για να κλείσετε τη φράση σας. Το μόνο που θέλω να πω, να σας ευχαριστήσω και να προσθέσω ότι στον τελευταίο κανονισμό για την ε, τιτλοποίηση φαίνεται όπως γίνεται με όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Υπάρχει το άρθρο 114 επίσης για τη συνθήκη, τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βλέπουμε στην ίδια γραμμή που είναι και άλλες αναφορές ότι τελικά δεν δίνουμε και πολύ σημασία στην προστασία των καταναλωτών και στα θεμελιώδη δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Τίποτα άλλο. Λυπάμαι που μίλησα τόσο πολύ. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τους αναφέροντες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις ε, πολιτικές ομάδες, οπότε θα αφήσουμε ανοιχτή την ανηφορά αυτή. Το ΕΛΚ βέβαια ε, είπε ότι θα μπορούσε να πάει το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή. Μα έτσι κι αλλιώ είχε απαντήσει, ναι, είναι αρμόδιοι για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν χρειάζεται να ζητήσουμε και πάλι έκθεση από την ε, γνωμοδότηση από την Οικονομική Επιτροπή. Αλλά η κυρία Κίρτον, η συντονίστρια, ζήτησε να αποφασίσουμε σε μια συνεδρίαση των συντονιστών μια μελέτη για την προστασία των καταναλωτών όσον αφορά τα ανυπόθηκα δάνεια για να δούμε πώς εφαρμόζονται όλα τα μέτρα που έχουν να κάνουν με τα ανυπόθηκα δάνεια και ο κύριος Γιάρα και η κυρία Κυρτοντάλινγκ το υπενθύμησαν ότι είχαμε πολλές αναφορές για τέτοια ζητήματα και όχι μόνο από την Ισπανία αλλά και από άλλες χώρες. Να δούμε πώς πρέπει να τροποποιηθεί η νομοθεσία. Και επίσης θα στέλναμε και επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών της Ισπανίας προκειμένου να ενημερωθούμε για τον νέο κανονισμό που ισχύει από 1η Νοεμβρίου του 2019, 2017-24 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του Δεκεμβρίου του 2017, που θέτει ένα γενικό πλαίσιο για την τιτλοποίηση και ένα ειδικό πλαίσιο για την απλή τιτλοποίηση, ώστε οι Ισπανικές αρχές να μας απαντήσουν την επιστολή αυτή και να μας εξηγήσουν τι άλλο χρειάζεται για να εφαρμοστεί πια αυτό το πλαίσιο και στην Ισπανία. Οπότε την αφήνουμε ανοιχτή. Ο κύριο Γιάρο όμω θέλει κάτι να προσθέσει. Αυτή είναι η πρόταση από πλευρά του Προεδρείου πάντω. Ναι, ναι, πολύ σωστά. Ε, συμφωνώ ε, με αυτό που λέτε, είναι σωστό. Αλλά να προσθέσω και κάτι, κυρία Πρόεδρε. Θα μπορούσαμε ίσως να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει κατά πόσο σκοπεύει να αλλάξει ή να προσαρμόσει την οδηγία για τα ανυπόθηκα δάνεια. Τώρα με τη νέα επιτροπή υπάρχει μια νέα ευκαιρία. Προς το παρόν έχουν πει ότι δεν πιστεύουν ότι είναι τέλεια. Ωραία για την μελέτη που προτείνεται, καλώς, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή που έχει το δικαίωμα πρωτοβουλίας. Οπότε νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να πει ότι όπως είπε λίγο πολύ, ότι ό,τι έχουμε τώρα δεν είναι τόσο τέλειο, οπότε ίσως θα πρέπει να αλλάξει. Για μένα είναι σαφές ότι υπάρχει τέτοια παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και θα ήθελα να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν σκοπεύει να αλλάξει. Βλέπω να γνέφει καταφατικά, οπότε υποθέτω πως ναι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να απαντήσει κάτι. Ναι, ναι, ναι. Όντω, θα αναθεωρήσουμε έτσι κι αλλιώ την οδηγία, γιατί υπάρχει μια ρήτρα αναθεώρηση στην οδηγία. Τώρα αν θα αναθεωρήσουμε και άλλα θέματα, αυτό εξαρτάται από την αξιολόγηση που θα κάνουμε. Πρόεδρος, καλώς. Ωραία. Ε, ακούσαμε τη ζήτηση το ΕΛΚΑ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απάντησε η Επιτροπή. Πρόταση της Πρόεδρου είναι να μείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή να συζητήσουμε τους συντονιστές ε, να προκειμένου να ετοιμάσουν μια έκθεση για αυτό το θέμα. Τρίτον, να ενημερώσουμε από την Επιτροπή Αναφορών την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα που έχει η νέα θητεία. μήπω σκοπεύει να τροποποιήσει, να αναθεωρήσει την οδηγία για τα ανυπόθηκα δάνεια. Και τέταρτον, να στείλουμε επιστολή στις Ισπανικές Αρχές το Υπουργείο Εθνική Οικονομία, ώστε να ενημερωθεί η Επιτροπή μα για το πώ εφαρμόζεται ο κανονισμό που ανέφερα πριν και η οδηγία για τα ενυπόθηκα δάνεια. Ευχαριστώ πολύ τους αναφέροντες πάντως που ήρθαν σήμερα. Σας ευχαριστούμε. Και συνεχίζουμε και περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι το σημείο 6 στην ημερήσια διάταξη. Είναι η αναφορά 91 κάθετος 2013 του κυρίου Σέρζ Γκράς, γαλλικής ηθαγένειας, εξ ονόματος της οργάνωσης για τη διαφάνεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Νομίζω όμως ότι δεν είναι εδώ αναφέρον, σωστά. Οπότε, θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Ματέο Σάλτο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχουν νέα στοιχεία για την αναφορά αυτή σε σχέση με ό,τι είχαμε μέχρι το 2014, οπότε δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Πρόεδρος, ωραία. Συντονιστές, κάποιος. Ο κύριος Γιάρ μήπως, κάποιος άλλος, κύριε Κίρτον. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, νομίζω ότι μπορούμε να την κλείσουμε αυτή την αναφορά. Δεν ξέρω τι λένε και οι συνάδελφοι. Η κυρία Κίρτον, Ντάρλινγκ. Εγώ δεν ξέρω τι να πω. Δεν έχω άποψη. Φαίνεται ότι υπάρχει μια επιστολή όμως που πήγε το 2018 στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και δεν ξέρω, είχαμε απάντηση. Α. Και στην απάντηση δεν υπήρξε τίποτα που να οδηγεί σε κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ε, τότε ναι, να συμφωνήσω κι εγώ ότι πρέπει να την κλείσουμε γιατί δεν βλέπω τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Πρόεδρος, ωραία, ακούσαμε τις πολιτικές ομάδες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεπώς, κλείνουμε την ε, αναφορά αυτή. Και περνάμε στο επόμενο σημείο, που το σημείο 7. Αναφορά 1721 του 2014 του Τάκη Χατζηγεωργίου, Κυπριακή Ιθαγένεια, σχετικά με τα εξαιρετικά υψηλά επιτόκια που χρεώνουν οι τράπεζε οι οποίε λειτουργούν στην Κύπρο. Δεν είναι όμως εδώ ο αναφέρον. Οπότε θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Μάρκα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Όσον αφορά την απάντηση που έχουμε ήδη δώσει, η νομική κατάσταση δεν έχει αλλάξει εξού και δεν έχω να πω τίποτε από αυτού. Πάντως, από την οικονομική άποψη βλέπουμε ότι αναφέρεται στις υποθήκες στην Κύπρο αναφέρον, οι οποίες έχουν μειωθεί πολύ τα επιτόκια δηλαδή, και είναι σήμερα στο ίδιο επίπεδο με τα γερμανικά. Όλοι γνωρίζουν ότι η αύξηση των τελών έχει να κάνει και με το κόστος του χρήματος, ε, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζονται συγκεκριμένοι ισολογισμοί που επηρεάζονται από τα μίξη υπηρετούμενα δάνεια. Έπειτα παίζει ρόλο ο ανταγωνισμός, το επίπεδο του ανταγωνισμού και η αξιολόγηση αντικτύπου που κάνουν οι τράπεζες όταν ε, παραχωρούν ένα δάνειο και εξαρτάται από την κατάσταση της οικονομίας, από τις εγγύησεις κλπ. Από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάντως εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο ανταγωνισμού στις χώρες μέλη. και να αυξήσουμε και την ε, δυνατότητα ε, πληρωμής των δανειοληπτών. Από ό,τι φαίνεται η κατάσταση σήμερα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν ε, όταν ετοιμάστηκε η αναφορά αυτή. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Πίτερ Γιάρ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρκεί. Είναι απόλυτα κατανοητό. Και έχουμε και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και προσπαθούμε να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να υπάρχει περισσότερος ανταγωνισμός. Κάτι έχει γίνει. Έχουν υπάρξει διακυμάνσεις στα επιτόκια, 2 με 15% είχαμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω ότι απάντησε, ότι είδαμε να υπάρχουν αποτελέσματα από την πολιτική ανταγωνισμού. Μπορούμε επίσης να πούμε ότι η Κύπρος είναι η χώρα που μας ενδιαφέρει σε αυτή την περίπτωση και είναι η Κύπρος η ίδια η οποία πρέπει να ασχοληθεί παρετέρω με αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε την αναφορά αυτή γιατί δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τον αναφέροντα. Αν υπάρχουν δυσκολίες πρέπει σε εθνικό επίπεδο να γίνουν προσφυγές. Εμείς, η Ombudsman, ε, ο Ευρωπαίος δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει τίποτα στην Κύπρο ίσως. Πάντως έχει πετύχει ε, μέχρι τώρα η κατάσταση και τα επιτόκια βρίσκονται σε νορμάλ κατάσταση πια και στην Κύπρο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ωραία, ακούσαμε την Επιτροπή, ακούσαμε και τις πολιτικές ομάδες. Έχουμε διαβάσει και την αναφορά. Την κλείνουμε λοιπόν. Έτσι, τι λέτε. Συμφωνείτε. Ωραία. Κλείνει. Και περνάμε στην επόμενη αναφορά που είναι η 0942 του 2018 του κύριου Μέρφυ, Βρετανική Σταγέννηση, εξ ονόματο των νέων Ευρωπαίων Φεντεραλιστών, σχετικά με τη θέσπιση κοινή Ευρωπαϊκή δημοσιονομικής πολιτικής. Ο αναφέρον δεν είναι εδώ, έτσι, σωστά. Οπότε θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Λουθία Πιάνα, που είναι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, θα μιλήσω αγγλικά. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο και τα μέλη. Η αναφορά έχει κάποια αξία για τον μηχανισμό σταθεροποίησης του, ε, της Ευρωζώνης Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει πρόταση για ευρωπαϊκό κανονισμό και για, τον, για τη διευκόλυνση της σταθεροποίησης ε, της ε, Ευρωζώνης, όμως ως προς τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και για την τελική σας σύσταση και την τοποθέτησή σας, οι εξελίξεις στο Συμβούλιο δεν πάνε παραδείγματος στην κατεύθυνση που θα ήθελε ο αναφέρον και κάποια από τα μέλη του Κοινοβουλίου. Ιδίω ε, ο προπολογισμό τη Ευρωζώνη δεν είναι κάτι που προβλέπεται για το άμεσο μέλλον, διότι υπάρχει το δημοσιονομικό εργαλείο για τη σύγκληση και την ανταγωνιστικότητα, αλλά δεν προβλέπεται να καλύπτει και θέματα σταθεροποίηση. Η συζήτηση για το μηχανισμό λοιπόν σταθεροποίηση δεν ξεκίνησε καν λόγω των διαφορετικών τοποθετήσεων των κρατών μελών. Η σταθεροποίηση είναι κάτι σαν ταμπού για κάποιους. Και για τον ε, ενοποιημένο εταιρικό φόρο που βλέπω να αναφέρεται στη σύστασή σας είναι μια μελλοντική εξέλιξη οι συζητήσει συνεχίζονται, όμως υπάρχουν πολλοί φραγμοί στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Οι συντονιστές τώρα. παρακαλώ. Κύριος Φλόρε. Κύριος Μάριο Φλόρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα στους συναδέλφους και τον αναφέροντα. Παίρνω το λόγο διότι ως μέλος του κινήματος των πέντε αστέρων και ως εκλεγμένος από τον Ιταλικό λαό δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν υπάρχει μια κοινή, οικονομική, μια κοινή νομισματική και οικονομική πολιτική δημοσιονομική και, και ε, νομισματική πολιτική που να καλύπτει όλα τα κράτη-μέλη. Αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μα υποχρεώνουν να σκεφτούμε κάποια πράγματα και όχι απλώ τα εκλογικά παιχνίδια και συμφέροντα που αντιμετωπίζουν τα οικονομικά συμφέροντα όπω τον καθένα βολεύει, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε του κοινά προβλήματα και τι κοινέ δυσκολίε. Θα πρέπει οι ευρωπαϊκοί λαοί να μην ε, αναγκάζονται μόνο να υποστούν στο πετσί του τι αποφάσει τη ε, Ευρωζώνη και η Ένωση να είναι μια πραγματική Ένωση όπου να μοιραζόμαστε και τα ωφέλη και τι επιτυχίε. Μετά τη συνθήκη του Μάστριχ, οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Νομισματική Ένωση είναι ακόμα εμιτελής, δημιουργώντας πολλούς κινδύνους και απειλέ για την Ευρωζώνη που μπορούν λόγω εσωτερικών ε, τριγμών να αντιμετωπίσουν προβλήματα και βεβαίως αυτό να, χτυπεί, να πλήξει τι βασικέ υπηρεσίε προ του πολίτε, όπω τι συντάξει, τα υγειονομικά και την ε, κοινωνική κάλυψη. Γι' αυτό λοιπόν συντάσσομαι με τον, ε, εμ, συμπαρατάσσομαι με τον αναφέροντα που όπως και η έκθεση των ε, πέντε συμπροέδρων ζητά να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ολοκλήρωση της δημοσιονομικής και, και νομισματικής πολιτικής με κοινέ αποφάσεις, ένα κοινό προπολογισμό και χωρίς βεβαίως να πλήττεται η εθνική κυριαρχία του κάθε κάτω μέλος, αλλά όπου θα πρέπει να γίνονται σεβαστές αρχές της συνταγματικότητας και της δημοκρατίας. Για να αντιμετωπίσουμε λοιπόν και το πρόβλημα των ε, φορολογικών παραδείσων, θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια ε, δημοσιονομική και κοινομισματική ένωση που να ε, επιτρέψει την ανακατανομή των κερδών που θα έχουμε από αυτήν την εφαρμογή. Ο κύριος Γιάρ, ευχαριστώ. Νομίζω η αναφορά μπορεί να μείνει ανοιχτή, διότι είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα και η όλη πολιτική διαδικασία έχει μέλλον εδώ έχουμε να κάνουμε μια σχετική αλαζονία των κρατών μελών που όλοι την εκδηλώνουν με τον ίδιο τρόπο. Θα πρέπει να μην βάζουν οι μεν εμπόδια στους δε. Το είδαμε και με την οικονομική κρίση, με τα κριτήρια για τη σταθεροποίηση της Ευρωζώνης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει εντοπίσει ότι κάποια κράτη-μέλη δεν έχουν προσφέρει τα απαραίτητα δεδομένα και στοιχεία για να κριθεί το κατά πόσον σεβάστηκαν τα κριτήρια. Υπάρχουν λοιπόν παραβιάσεις στο σύστημα του ευρώ και της ευρωζώνης και εάν υπάρξει μια περαιτέρω κρίση θα αντιμετωπιστούν παρόμοια προβλήματα. Η αλαζονία λοιπόν των κρατών μελών μέσα από τις εθνικές τους βουλές, το ξέρω ας πούμε από την Γερμανία, όπου είναι υποχρεωμένοι οι αρμόδιοι φορείς της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης να δίνουν τα σχετικά στοιχεία και δεδομένα Οπότε θα έλεγα ότι η συγκεκριμένη αναφορά θέτει μια συζήτηση κέρια σημασία, την οποία δεν θα, θα πρέπει να την κλείσουμε, αλλά να τη συνεχίσουμε. Το Κοινοβούλιο μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δει την, ε, τις ε, αναγκαίες αλλαγές και να τις προτείνει στα κράτη-μέλη που μπορεί απλώ να λαμβάνουν γνώση προ στιγμή, αλλά εγώ την αναφορά δεν θα την έκλεινα, γιατί θα ήταν καλό η συζήτηση αυτή να συνεχιστεί. Μπορεί να χρειαστούν αρκετά χρόνια, αλλά δεν θα έλεγα ότι πρέπει να μπει στο χρονοτούλαπο ε, το όλο θέμα. διότι διαρκώς μόλις προκύψει μια νέα κρίση όλοι ξεχνάνε τα, τους κανόνες και τα ε, ισχύοντα και κοιτάζουν απλώς πώς μπορούν να διασώσουν την κατάσταση. Ευχαριστούμε κυρία Κίλτον Ντάρλι. Πολύ σύντομα, ε, συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Γιάρ. Ε, υπάρχει ομοφωνία εδώ στην Επιτροπή. Όμως από την πλευρά των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών όντως είναι ένα σημαντικό ζήτημα και η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι η συζήτηση είναι παθιασμένη και μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο σημαντικό είναι η αναφορά να παραμείνει ανοιχτή. Και καλό θα είναι να την αναπέμψουμε και στην αρμόδια επιτροπή. Ελπίζουμε ότι θα γίνει και κάποια κίνηση στο Συμβούλιο προς μια πολιτική με περισσότερη ελεγγύη στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις πολιτικές ομάδες και αποφασίζουμε να παραμείνει ανοιχτή. Ζητάμε γραπτή ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως είπαμε γιατί δεν έχουμε γραπτά ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. και θα ζητήσουμε γνωμοδότηση από την ε, Οικονομική Επιτροπή. Εντάξει, ωραία. Και συνεχίζουμε και περνάμε στο επόμενο σημείο της υπηρεσίας διάταξης, 9, που είναι η αναφορά 0645-2017 του Μάρκ Σμέτς, Βελγικής Ιταγέννης, σχετικά με τον φερόμενο σταθέμητο ανταγωνισμό στην αγορά ίνων κοινοπνευματοδών του Βελγίου λόγω της αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Είναι εδώ ο κύριος Σμέτς. Ναι. Πέντε λεπτά έχετε στη διάθεσή σας, παρακαλώ, για να μας παρουσιάσετε την αναφορά σας. Κύριε Σμέτ, παρακαλώ. Ή δεν είναι εδώ. Α, δεν είναι εδώ. Οπότε τότε θα δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που είμαι εδώ και μπορώ να σας παρουσιάσω την απόκριση Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην αναφορά αυτή, η οποία σχετίζεται, όπως ξέρετε, στις ε, συνεχείς αυξήσεις των ειδικών φορών κατανάλωσης από το Βέλγιο, που επηρεάζουν ε, μικρούς ε, πολιτές υνοπνευματοδών στο Βέλγιο, γιατί μπορούν οι καταναλωτές να αγοράσουν πνευματόδη σε άλλα κράτη-μέλη, το οποίο δημιουργεί αθέμητο ανταγωνισμό λόγω της κατάχρησης που γίνεται του δικαιώματος αγοράς νοπνευματοδών σε χώρες με μικρότερους ειδικού φόρους κατανάλωσης. Αυτό υπάρχει, αλλά οι κανόνες ε, που διέπουν την αγορά αυτή όντως έχουν κάποια προβλήματα. Ο ελάχιστος φόρος ε, αυτός για τα ενοπνευματόδη βρίσκεται στην 9284 μια οδηγία η οποία εγκρίθηκε το 92 με την εκκίνηση της ενιαίας αγοράς υπόκειται στους κανόνες της ε, ειδικέ νομοθετικές διαδικασίες δηλαδή ψηφοφορία ομόφωνη στο Συμβούλιο. Και επιπλέον η νομοθεσία πλαίσιο που καλύπτει την ε, οδηγία αυτή θέτει ελάχιστους εναρμονισμένους, ε, εναρμονισμένες ε, τιμές και όχι ανώτατες, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί ο καθένας να θεσπίζει ειδικούς φόρους κατανάλωσης υψηλότερους από τα χαμηλότερα αυτά κατόφλια που μπορεί να φτάσουν και σε πολύ ψηλά ποσά για τα ενοπνευματόδη για να ανταποκριθούμε στην αναφορά αυτή για την εναρμόνιση των κανόνων. Εμείς προσπαθήσαμε ε, αυτούς τους ελάχιστους συντελεστές να τους αυξήσουμε σε πιο ρεαλιστικούς σε σχέση με αυτό που θεσπίθηκε το 1992, γιατί βέβαια ε, εδώ έχουμε το θέμα της τιμεριθμικής αναπροσαρμογής που δεν είχε γίνει. Κάναμε μια πρόταση το 2006 και ενώ στηρίχθηκε από μεγάλο αριθμό κρατών μελών, η πρόταση αυτή δεν κατάφερε να βρει ε, την ομοφωνία, γιατί κάποια κράτη-μέλη λόγω εθνικών ε, θεμάτων δεν στήριξαν την πρόταση αυτή. Εμείς αποσύραμε το 2015 την πρόταση γιατί ε, ήταν στο τραπέζι για όλα αυτά τα χρόνια γιατί δεν είχαμε καμία εξέλιξη ή πραγματική σύγκληση μεταξύ κρατών μελών για θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής, για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα ενωπνευματώδη. Και κατανοούμε πως έκτοτε δεν έχει αλλάξει αυτό για τον αθέμητο ανταγωνισμό λόγω της κατάχρησης του της δυνατότητας αγοράς σε άλλα κράτη-μέλη. Το, δι... το Δεκέμβριο του 2017 το Συμβούλιο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, δει το θέμα των εξαποστάσεων αγορών από μεμονωμένα άτομα ε, ενοπνευματοδών ποτών όπως επίσης και από ε, γενικά καταστήματα εκτός συνόρων και προσπαθήσαμε να μειώσουμε αυτούς τους δασμούς ε, γιατί είχαμε περιπτώσεις ατόμων που επικαλέστηκαν προσωπική κατανάλωση για να μεταπολίσουν μετά αυτά τα ενοπνευματόδη. Τον Οκτώβριο του 2017 κάναμε μία μελέτη για τα άρθρα 32 και 36 της οδηγίας που λήπτη τις ε, γενικές διευθετήσεις για τους εναρμονισμένους ειδικού φόρους κατανάλωσης και ε, τη στιγμή που η μελέτη αυτή ε, πρόκειται να ε, περατωθεί θα τη στείλουμε στη Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις. Βέβαια, αναγνωρίζουμε τις ανησυχίες όλων των εμπλεκομένων και του αναφερόμενου που ζήτησε να ε, συνεισφέρει στην έκθεση αυτή, στη μελέτη αυτή. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι οι ενδεχόμενες μελλοντικέ προτάσεις. Γνωρίζετε όλοι πως αυτή τη στιγμή η τρέχουσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη σύνθεσή της ε, απλώς ε, εκτελεί υπηρεσιακά καθήκοντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν οι πολιτικές ομάδες θέλουν να πάρουν το λόγο. Όχι. Ναι, αν και έχουμε εσωτερική αγορά, και υπάρχουν και ευθύνε των κρατών μελών. Μελικοί μπορούν να αυξήσουν τους ειδικού φόρους, πράγμα που επιτρέπεται. Η εναρμόνιση δεν έχει γίνει αποδεκτή. Υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί βεβαίω ε, στο εμπόριο λόγω της εσωτερικής αγοράς. Σε κάποιους δεν αρέσει αυτό και θα έπρεπε να υπάρχει κατά την άποψή τους εναρμόνιση των ειδικών φόρων. Κοιτάζω τώρα τους, τη συνάδελφο Διότι και οι δύο αποφάσει θα μπορούσαν να αιτιολογηθούν, είτε να την αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά, είτε να την κλείσουμε. Είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών σε κάθε περίπτωση να αυξήσουν, να μειώσουν του εθνικού φόρου εφόσον τα επιθυμούν. Εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμη κοιτάζει κατά πόσον θα μπορούσε να υπάρξει ένα καλύτερο επίπεδο εναρμόνιση. Το θέμα είναι τι μπορεί να αποφασίσει και η Πρόεδρο. σω αποφασίσετε εσεί η ίδια, κυρία Πρόεδρε. Αφήνουμε εσά να αποφασίσουμε, να λάβετε την απόφαση εμείς, μπορούμε να δεχτούμε και τις δύο εναλλακτικέ, είτε να μείνει ανοιχτή είτε να κλείσει. Πάντως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα αυτό να, να, να της πούμε ότι θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε. Ευχαριστώ. Συμφωνώ. Είναι το είδος της αναφοράς όπου υπάρχει ένα ε, ελάχιστο επίπεδο φόρων και οι χώρες αποκλίνουν διότι έχουν αρμοδιότητα. Ε, για κάποιους έχει αρνητικό αντίκτυπο στον τομέα που δραστηριοποιούνται και πλήττει εν μέρη τα συμφέροντά τους, αλλά εμένα μου αρκούσε η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βρίσκω πολύ θετικό το γεγονός ότι οι αναφέροντες έχουν άμεση εμπλοκή στην όλη εξέλιξη και στις διαπραγματεύσεις, οπότε από αυτήν την έννοια νομίζω ότι είναι λογικό να κλείσει η ανάφορα. Εάν χρειαστεί στο μέλλον, οι αναφέροντες μπορούν και πάλι να υποβάλουν νέα αναφορά και να ζητήσουν και πάλι την δική μας την υποστήριξη. Όμως στο πλαίσιο της συγκεκριμένη αναφοράς, <clears throat> οι πολιτικοί ηθήνοντες έχουν νομίζω αποταθεί απευθεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η άποψή τους έχει εισακουστεί. Η Βελγική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και οι Βελγικές Αρχές γνωρίζουν, οπότε μπορούν να επιληφθούν εφόσον το θέλουν. Ευχαριστώ. Ε, οι συντονιστές συμφωνούν λοιπόν, οπότε κλείνουμε την αναφορά αυτή. Περνάμε στο σημείο 10, αναφορά 1190 του 18 του Γκρεγκουάρ Σερβέ, γαλλική σχετικά με του φόρου επί των εισαγωγών ηλεκτρικών ποδηλάτων από την Κίνα. Δεν είναι εδώ αναφέρον, οπότε θα δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον κύριο Χάρλ Σμιτ. Ευχαριστώ η αναφορά έχει να κάνει με, την, ε, ε, με τους κανόνες για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα από την Κίνα και την, ε, των ηλεκτρικών δηλαδή από την Κίνα και τους κανόνες αντι-dumping. Δύο είναι τα βασικά σημεία που ήθελα να θίξω. Πρώτα απ' όλα τι έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά γιατί το έκανε οι κανονες αντι anti-dumping υπογραμμώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κοιτάξει τι γίνεται με τα ηλεκτρικά ποδήλατα από την Κίνα. Όμως οι σχετικές επιχειρήσεις και η παραγωγή, η εισαγωγή, η εξαγωγή και οι πολιτές των ηλεκτρικών ποδηλάτων είχαν τη δυνατότητα να απαντήσουν και να δούμε τι γίνεται με την συγκεκριμένη υπόθεση. Η έρευνά μας έδειξε ότι τα κινέζικα ηλεκτρικά ποδήλατα δεν ε, πλήττουν την, ε, τους κανόνες αντι-dumping. Μάλλον πλήττουν τους κανόνες αντι-dumping και προ, επιβάλλουν, προξενούν ζημιές, οικονομικές ζημιές στις ευρωπαϊκές εταιρείες το θέμα είναι ότι ο σχετικός κλάδος παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιδοτείται και θα πρέπει να αναγνωριστούν αυτά και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Τα κανονικά ποδήλατα χωρίς ηλεκτρικό κινητήρα ε, δεν, ε, μάλλον έχουν ειδικού κανόνες εισαγωγή και είναι πολύ περιορισμένα, οπότε τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν όπως χρησιμοποιούνται και για τα ευρωπαϊκά ποδήλατα. Είναι σημαντική η παραγωγή των ποδηλάτων για το θέμα της κινητικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ή άλλως. Μιλάμε για μια αγορά με πολλά εκατομμύρια οδηγούς ποδηλάτων Οπότε είναι ένα σημαντικό, ε, ένα κλάδος που, που υποστηρίζει το σχέδιο του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ η κυρία Κίτον πρώτα. Ε. Ναι. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η δικιά μου εμπειρία σε θέματα διεθνούς εμπορίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ότι για να φτάσει η Επιτροπή να εφαρμόσει την αντι-dumping έχει ε, προβεί σε μελέτες αντικτύπου ενδελεχώς ε, και έχει ήδη διαμαρτυρηθεί για, τα, ε, για το dumping το οποίο διαπιστώνει όπως είπε και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε η κάθε περίπτωση βέβαια μπορεί να είναι διαφορετική πάντα κάποιος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πλήττεται αρνητικά. Δεν είναι τα πράγματα άσπρο-μαύρο. Πάντως, για να είμαστε δίκοι, καλό θα ήταν να αφήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά ακόμα, ώστε να επιτρέψουμε να εξεταστεί περισσότερο και να δούμε αυτά τα μέτρα που έχει εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς θα προχωρήσουμε το χρόνο, τι επιπτώσεις θα έχουν όσο περνάει ο καιρός, μήπως κάποια στιγμή χρειαστεί να μετριαθούν ή να αλλάξουν. Είναι σαφές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τα μέτρα αντι-dumping είναι δίκαια και σωστά. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πλήττονται από αυτά. Γι' αυτό λέω να παραμείνει ανοιχτή αναφορά. Και αν υπάρχει κάτι νέο από πλευράς του αναφέροντος, θα έχουμε έτσι την ευκαιρία να κάνουμε ξανά τη συζήτηση στα πλαίσια της νέας συγκυρίας. Ο κύριος Γιάρ. Δεν θέλω να αλλάξω την ε, συμφωνία μεταξύ μας, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι τα μελέτησε διεξοδικά, ότι κοίταξε τα μέτρα και τα εφήρμοσε. Οπότε πιστεύω ότι η αναφορά θα μπορούσε και να κλείσει με βάση αυτήν την εξήγηση. Η όλη η διαδικασία συνήθω κρατάει τόσο πολύ Τώρα κάπου έχουμε φτάσει και μπορεί κάτι να γίνει. Εάν λοιπόν κατάλαβα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σωστά, τα μέτρα αντι-dumping έχουν εφαρμοστεί. Μπορεί να κλείσει η αναφορά. Και εφόσον υπάρξει μελλοντικά κάποιο πρόβλημα, μπορεί ο αναφέρον να ξαναυποβάλει μια αναφορά. Εάν, εφόσον όλα έχουν ήδη εφαρμοστεί, μπορεί ήδη να κλείσει η αναφορά. Εάν πείτε ναι, θα τα βρούμε. Η αρμονία και η συμφωνία είναι πάντοτε καλό πράγμα, αλλά εφόσον υπήρξαν μέτρα θα πει ότι προηγήθηκε διεξοδική έρευνα. Τα μέτρα την dumping επιτρέπουν ίσω κάνω στο παιχνίδι σίγουρα, αλλά υπάρχουν και εταιρείε ενδεχομένω στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν ε, πληγεί ε, ήδη. Εάν κλείσει λοιπόν η αναφορά, η σύστασή μου θα ήταν κλείνοντα και ενημερώνοντα τον αναφέροντα ότι την κλείνουμε, να αφήσουμε τη δυνατότητα, εάν θελήσουν οι αναφέροντε, να υποβάλουν νέα αναφορά. Εάν τα πράγματα αλλάξουν, πάρουν άλλη τροπή, και αναγνωρίζοντας ότι οι κανόνες αντι-dumping πρέπει να ισχύουν διαρκώς. Και ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν ισότιμοι κανόνες ανταγωνισμού σε σχέση με τους Κινέζους που εξάγουν τα ποδήλατά τους, οπότε δεν θα προκύψει και κάτι ανάλογο στο μέλλον. Αυτό θα θέλαμε να αποφευθεί. Και εμένα πολύ μου αρέσει η αρμονία. Ωραία, χαίρομαι που πετύχατε την αρμονία ο κύριος Γιάννη και η κυρία Ήττον. Θα συνεχίσουμε γιατί εμένα μου άρεσε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, γραπτά αναφέρθηκε στη δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσει προσωρινή επανεκτίμηση, για παράδειγμα μετά από ένα χρόνο μετά τη λήξη της τρέχους απόφασης κατά του ντάμπινγκ. Γιατί αν δεν δώσει στον αναφερόμενο τη δυνατότητα να ζητήσει κάτι τέτοιο, δηλαδή αξιολόγηση προσωρινή ε, μετά από ένα χρόνο κτλ. Ε, θα λειτουργήσει. Είτε κλείσουμε την αναφορά ή την αφήσουμε ανοιχτή. Ας την αφήσουμε λοιπόν ανοιχτή γιατί αν σε ένα, αφού πέρασε ένας χρόνος δεν... Ε, Α, να δούμε λοιπόν σε ένα χρόνο. Αν δεν λάβουμε αντίστοιχη αναφορά με στον επόμενο χρόνο και αν δεν επανέλθει ο αναφερόμενος, να κλείσει αυτόματα τότε. Έτσι ώστε να πετύχουμε την αρμονία ανάμεσά μας. Ωραία, αυτό θα κάνουμε. Να περάσουμε λοιπόν στην επόμενη, την οποία έχει ζητήσει ο Σέρς Λεκουέ από τη Γαλλία. Είναι η 1190-2018. Α, είναι η επόμενη, είναι η 0328 ε, για ε, τους ε, ε, περιφερειακούς ε, αλληλέγγυους της Βρετάνης με 12 υπογραφές για την έκθεση των εργαζόμενων στα αγροκτήματα σε ε, ζυζανιοκτώνα. Ήθελα να σας ρωτήσω, θα πάρετε το λόγο όλοι ή ένας, γιατί είναι 5 λεπτά, άρα τότε θα έχετε από 2,5 λεπτά. Και μετά στο κλείσιμο θα σας δώσουμε άλλα 2 λεπτά, ένα και ένα ή ένα άτομο για 2 λεπτά. Οπότε, εσείς είστε ο κύριος Λεϊκού. Μπορείτε να ξεκινήσετε εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλαμε να ακούσουμε μια απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι η τρίτη φορά που ερχόμαστε για την ε, προστασία αυτή των εργαζόμενων. Να σας πω πως περιμέναμε και την απάντηση του σχετικού αρμοδίου γαλλικού Υπουργείου και θέλουμε ε, πριν συνεχίσουμε εμείς να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί πιστεύω ότι έχει εξελίξει και πρέπει να ενημερωθούμε. Ωραία. Ωραία. Θα σας ξαναδώσω το λόγο μετά και θα σας αφήσω να μιλήσετε πέντε λεπτά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Γκρίφιθς. Για να σας ενημερώσω λοιπόν για τα θέματα αυτά την τελευταία φορά που τα συζητήσαμε, τον Απρίλιο αν δεν κάνω λάθος με την αναφορά αυτή, να σας πω πως τα θέματα που έθεσαν οι αναφερόμενοι έχουν να κάνουν και με την προστασία των εργαζομένων και την προστασία των προϊόντων. Οπότε έχω και συνάδελφο από την DG Employment εδώ για την ασφάλεια των εργαζομένων. Τρία θέλω να πω Πρώτα απ' όλα την έκθεση ε, ελέγχου για τη Γαλλία για τη βιώσιμη χρήση ζυζανιοκτώνων έχει δημοσιευθεί στη Γενική Διεύθυνση Σάντες στη σχετική, στο σχετικό ιστότοπο με την απάντηση των γαλλικών αρχών. Μετά λοιπόν από την αλληλογραφία που είχαμε ένα σχέδιο δράσης εστάλει από τη Γαλλία για τα γενικότερα θέματα της βιώσιμης ε, χρήσης ζυζανιοκτώνων και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα και το 2020 έτσι ώστε να εφαρμοστούν όπως μας έχουν υποσχεθεί για τα συγκεκριμένα θέματα της αναφοράς για την ασφάλεια των εργαζομένων στη Βρετάνη. Εδώ περιμένουμε την απάντηση των γαλλικών αρχών. Από την τελευταία συζήτηση λοιπόν λάβαμε μία απόκριση από την την Αρμόδια Υπηρεσία για τα Εργασιακά. Στείλαμε και στο Υπουργείο Γεωργίας μια επιστολή ε, για ε, αποσαφηνίσεις γιατί είχαμε κάποια κενά. Καθυστέρησαν τρεις περίπου μήνες στο να μας στείλουν μια απάντηση. Αλλά τελικά η μόνιμη αντιπροσωπεία παρενέβη και έχουμε αυτή τη στιγμή μια ικανοποιητική απάντηση την οποία λάβαμε 17 Οκτωβρίου και η αρχική μας αξιολόγηση είναι πως δίνει τις ε, απαραίτητες πληροφορίες για να κλείσουμε εμείς την αξιολόγηση. Αν συμφωνήσετε λοιπόν θα το κάνουμε με γραπτή διαδικασία προς την Επιτροπή έτσι ώστε να σας καταθέσουμε τη σχετική σύνοψη. Θα δώσω το λόγο και στον ε, εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Employment, τον κύριο Εβελίν. Ευχαριστώ. Για το θέμα της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων που προέκυψε κατά την έρευνα που κάναμε για την αναφορά, ε, ευθυγραμμίζουμε απόλυτα με τα όσα είπε ο συνάδελφος, αξιολογούμε αυτή τη στιγμή τις προφορίες που έστειλαν οι γαλλικές αρχές για να δούμε αν συμμορφώνονται με τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πολλά ε, νομοθετήματα στην, ε, στο σχετικό χώρο θέτουν ελάχιστες ε, προδιαγραφές και τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν πιο αυστηρούς κανόνες και η εφαρμογή είναι στο μεγαλύτερο βαθμό αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και εμείς αξιολογούμε λοιπόν τις πληροφορίες που μας στείλανε. Όπως ακριβώς είπε ο συνάδελφο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα λοιπόν, ναι, θα δώσω το λόγο στον αναφερόμενο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι η Γαλλία σε επίπεδο δηλώσεων τα πάει πολύ καλά. Όμω στην πρακτική εφαρμογή των οδηγιών και των κανονισμών τη Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα ανάβησο μεταξύ των όσων δηλώνει και όσων πράττει. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε εδώ και κάποιου μήνε είναι ότι υπάρχει μια σωρία αποφάσεων από ε, πρωτοδικεία, από διοικητικά δικαστήρια, από ειρηνοδικεία και έχουμε φτάσει στο Συμβούλιο Επικρατείας που πλαισίωσε τη χρήση των στη Γαλλία μια οδηγία που ε, έχει αντικατασταθεί από εγκύκλιο του Υπουργείου Γεωργίας. Αυτό που ζητάμε λοιπόν εμείς ως αναφέροντες είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως έκανα με την πρώτη οδηγία, να αναλάβει δράση. Ε, και θα θέλαμε, εφόσον δεν υπάρχει αποκατάσταση, να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Ευχαριστούμε πολύ. Ο άλλος αναφέρον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε συνέχεια, ο συναδελφός μου, και ού, σήμερα από την προηγούμενη φορά που ήρθε εδώ, φαίνεται να έχουμε ένα σύνολο δεδομένων στα χέρια μας, τα οποία δεν είχαμε την προηγούμενη φορά. Λόγω χάρη, έχουμε έναν αριθμό ο οποίος πραγματικά σοκάρει και έχει συγκεντρώσει ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας των Γεωργών στη Γαλλία που έχει να κάνει και με τους χρήστες και τους ε, ε, ε, ασθενείς από τη χρήση φυτοφαρμάκων. Έχουμε 2.500 περιπτώσει νόσου Πάρκινσον στη Γαλλία που προκαλούνται από τη χρήση αυτών των φυτοφαρμάκων χωρί να μιλήσουμε για άλλες νόσους όπως η υπερευαισθησία στα χημικά ε, προϊόντα ή άλλες νευρολογικές ασθένειες, ή καρκίνων και που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν αναγνωρίζονται ως επαγγελματική ε, πάθηση. Ε, Παρατηρούμε, Πρόεδρε, αύξηση του αριθμού στον τομέα της χρήσης φυτοφαρμάκων στην Γεωργία. Πάνω από 11%. Κοιτάζουμε επίσης και βλέπουμε ότι υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη έκθεση των γειτόνων των χρηστών, διότι οι δοσολογίες ε, μειώνονται, αλλά ο αριθμός των ε, ε, ψεκασμών αυξάνεται. Αυτό, που σημαίνει αυτό σημαίνει ότι σήμερα ο γεωργικός πληθυσμός αλλά και των γειτόνων ε, είναι θύματα μεγαλύτερης έκθεσης. Δεν θα έπρεπε λοιπόν η διαδικασία αυτή να κλείσει. Πιστεύω ότι το καλύτερο είναι να μείνει ανοιχτή για να έχουμε τη δυνατότητα να ε, αναλάβουμε δράση και να ζητήσουμε την προστασία των θυμάτων ή να υπάρξουν αποζημιώσεις. Και πρέπει να πω ότι όταν οι γαλλικές αρχές δεν αναλαμβάνουν ε, τις ευθύνες τους και δεν προστατεύουν τους πολίτες, τότε πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξουν και διώσεις κατά των υπευθύνων. Η Γαλλία έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώνει στοιχεία και έχουμε τέτοια αριθμητικά στοιχεία στα χέρια μας, πραγματικά είναι... μας αφήνουν άφωνος. Ως γεωργός και κάτοικος της υπαίθρου ξέρω τα πολύ καλά την κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν ήρθαμε σήμερα εδώ να πούμε ότι θα πρέπει η χρήση των φυτοφαρμάκων να πάρει μια αντίστροφη πορεία. Διότι με τα φυτοφάρμακα έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που πραγματικά είναι ε, ανάλογη με τις διαστάσεις που είχε το πρόβλημα του αμοιάντου πριν κάποια χρόνια. Πράγμα που δεν επιτρέπεται. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Πολιτικές ομάδες τώρα. Παρακαλώ, κύριε Μέστρε. Ευχαριστώ πολύ. Ακούω, παρακολουθώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους αναφέροντες είναι ένα θέμα αναμφίβολα σημαντικό από κάθε άποψη και γι' αυτό και υπάρχουν και πάρα πολλές ευρωπαϊκές οδηγίες που ρυθμίζουν την χρήση των φυτοφαρμάκων αυτών είναι πολύ σημαντικό το πώς υποφέρουν οι άνθρωποι που πλήττονται από, τέτοια, από τέτοιες ουσίες. Άκουσα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζητούν εκθέσεις μετά από τρεις μήνες, αλλά τελικά οι πληροφορίες που έχουν ζητήσει από την γαλλική δίκηση δεν έχουν ολοκληρωθεί, δεν έχουν σταλεί. Οπότε σαφώς και πρέπει να μείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή μέχρι να διευκρινιστεί γιατί πρόκειται για την υγεία των ανθρώπων που βάλετε από τις ουσίες αυτές των φυτοφαρμάκων και να δούμε ποια είναι ακριβώς η σχέση και δεν πρόκειται μόνο για τους ανθρώπους, πρόκειται και για το περιβάλλον. Δεν είναι μόνο η δημόσια υγεία, είναι και το περιβάλλον πώς καταστρέφεται από το φαρμακό. Οπότε η γαλλική δίκηση δεν έχει στείλει ακόμα τις πληροφορίες που θα έπρεπε, οπότε πρέπει να συνεχίσουμε και να ζητάμε τις πληροφορίες αυτές. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ωραία, παρακαλώ, κύριε Πανέλη. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι σαφής η κατάσταση. Δεν υπάρχει καμιά αφιβολία ότι πρέπει να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά αυτή. Είναι προφανές από τις έρευνες που έχουν γίνει μέχρι τώρα ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό. Σοβαρό πρόβλημα. Και ίσως θα πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι πιο αποτελεσματική στις έρευνές της και να προχωράει και πιο γρήγορα, γιατί προς το παρόν κρατάει πάρα πολύ αυτή η υπόθεση. Υπάρχει ψηλό κίνδυνος εξαιτία των καθυστερήσεων αυτών. Έχουμε εδώ πέρα όλους τους ε, αναφέροντες μπροστά μας με τους πάρα πολύ σοβαρούς ε, και βάσιμους φόβους τους. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να πιέσουμε να προχωρήσει πιο γρήγορα αυτή η υπόθεση. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Για να ολοκληρώσουμε. Δύο λεπτά παρακαλώ να φέρω. Σε ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω ότι όλα υπόθηκαν. Εμείς διαπιστώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν δημοσιεύσει κείμενα όσον αφορά οδηγίες και κανονισμούς που είναι πραγματικά αξιοθαύμαστα κείμενα και προστατεύουν τον πληθυσμό και τους εργαζόμενους. Μετά είναι καθήκον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ελέγχει ε, το πώς εφαρμόζονται όλα αυτά τα κείμενα. Πολλές φορές έχει καταδικαστεί το γαλλικό κράτος από διάφορα δικαστήρια εξαιτία ε, του δράματος ε, που ζούμε. Εδώ οι τρεις που με συνοδεύουν έχουν δηλητηριαστεί και τρεις από φυτοφάρμακα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Αναφορών του θα πρέπει να πιέσουν τη γαλλική κυβέρνηση για να κινητοποιηθεί και να αναλάβει συγκεκριμένα μέτρα που όλοι ζητάμε. Παρακαλώ. Και εσείς. Ευχαριστώ. Ναι. Κοιτάξτε, επιτρέψτε μου και εμένα λίγα δευτερόλεπτα. Στόσο λέει η Γαλλία. Φαίνεται να υπάρχει βούληση να διαχωρίσει να διαχωρίσει εντελώ το θέμα της εμπορίας. Βλέπετε τα φυτοφάρμακα είναι προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας για τις επιχειρήσεις. Το εμπορικό σκέλος δηλαδή είναι σημαντικό. Και δεν υπάρχει βούληση μείωσης γιατί πρόκειται για μεγάλες επιχειρήσεις, μεγάλους συνεταιρισμούς κτλ. που έχουν συμφέρον να πουλάνε τέτοια προϊόντα επικίνδυνα. Αυτό λοιπόν που λείπει στις διατάξεις της Γαλλίας είναι το ότι θα έπρεπε συστηματικά η ρύθμιση με εναλλακτικές προτάσεις αντί για τη χρήση των συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων στη Γεωργία. Και όσο δεν θα υπάρχει αυτό, όσο δεν θα έχουμε πάει πιο μακριά δηλαδή για να προτείνουμε εναλλακτικές και έτσι να βοηθάμε τους ε, εμπόρους, δεν θα βοηθήσει πολύ και δεν πρόκειται να μειωθεί η χρήση των φυτοφαρμάκων αυτών. Πρόκειται για την υγεία τη δικιά μα, των παιδιών μα, των εγγόνων μα που διακυδεύεται εδώ. Το θέμα των φυτοφαρμάκων για μα είναι ένα αγώνα που πρέπει να κερδίσουμε. Είναι δυνατόν να έχουμε μια διαφορετική γεωργία αν χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που μπορούμε στη διάθεσή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους αναφέροντες. Ακούσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακούσαμε και τις, ε, τους βουλευτές από τις πολιτικές ομάδες, οπότε διατηρούμε ανοιχτή την αναφορά αυτή και ζητάμε από τις γαλλικές αρχές, θα στείλουμε υπενθύμηση μετά την πρώτη που στείλαμε στις γαλλικές αρχές μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας ώστε να ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών για την κατάσταση και για το πώς έχει προσαρμόσει τις ρυθμίσεις. Ευχαριστούμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να συνεχίσει να μας ενημερώνει με λεπτομερείς πληροφορίες. Σίγουρα και η ΕΝΒΗ δουλεύει πάνω σε αυτά. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μας ενημερώνει για τη συνέχεια που δίνεται γιατί πρέπει φυσικά να προστατεύουμε την υγεία όλων των Ευρωπαίων. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν και τους αναφέροντες που ήρθαν εδώ σήμερα. Συνεχίζουμε και περνάμε τώρα στο σημείο 12. Αναφορά 60 του 2017 ενός πολίτη γερμανικής ηθαγένειας με δύο υπογραφές σχετικά με τη μη επιβολή από τις γερμανικές αρχές του κανονισμού 1069 κάθετος του 2009 προς μια μη συμμορφούμενη κατάσταση βιαερίου στο Σουάμπι Hall. Δεν είναι εδώ ο αναφέρον, οπότε θα δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλμπερτ, από τη Σάντε. Madam Chair. Good afternoon. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Η αναφορά έχει να κάνει με την εγκατάσταση ε, μονάδας βιοαερίου στο Σφάμπσεσάλ και αναφέρον θεωρεί ότι η έγκριση, η έγκριση δόθηκε κατά παραβίαση του κανονισμού 1069-2009 για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων. Πριν την αναφορά αυτή, το 2017 ασχοληθήκαμε με μία προσφυγή παρόμοιου, παρόμοιας φύσης για τα ίδια γεγονότα και εξετάσαμε τότε εκείνη την ε, ε, προσφυγή και κλείσαμε την υπόθεση διότι επί της αρχής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερευνά έρευνας, ερευ, περιπτώσεις συστηματικής μη συμμόρφωσης όπου τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν τον ε, κοινοτικό νόμο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θεωρήθηκε ότι ήταν εκτός αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναλάβει δράση ή να αποτιμήσει την συγκεκριμένη υπόθεση και τις προεκτάσεις της. διότι έτσι θα πληττετώ η ε, κατανομή αρμοδιότητα μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κράτων μελών και τη σωστή εφαρμογή της κοινωτικής νομοθεσίας. Όμως κατόπιν του αιτήματο ε, της Επιτροπής Αναφορών στις αρχές του 2019 για το θέμα αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε ε, επιστολή προς την Γερμανία τον Ιούλιο και ζήτησε από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές να συγκεντρώσουν περαιτέρω πληροφορίες για ενδεχόμενες μελλοντικέ δράσεις. Πρέπει να πω ότι δυστυχώς ω τώρα δεν έχουμε λάβει απάντηση από τους αρμόδιους γερμανικούς φορείς της γερμανικές αρχές. έχοντα διαπιστώσει ότι υπάρχουν περισσότερες περιπτώσεις παραβίασης, να θυμίσω ότι βάσει των σημερινών μας στοιχείων, στη βάση δεδομένων μας, έχουμε πάνω από 6.000 μονάδες βιοαερίου που έχουν εγκριθεί βάσει του κανονισμού για τη χρήση των ζωικών υποπροϊόντων στη Γερμανία και τουλάχιστον 800 από αυτές τις μονάδες βρίσκονται στη Βάτη ε, Βουτεμβέργη. Κάθε περίπτωση σφάλματος ή πλημελούς εφαρμογής των κανόνων είναι σίγουρα περιττή. Καταλαβαίνουμε την ε, αγανάκτηση των ε, αναφερόντων, όμως συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι αυτή η μεμονωμένη περίπτωση πρέπει να εξεταστεί από τις αρμόδιες αρχές στο συγκεκριμένο κρατήδιο στη Γερμανία ή τέλο πάντων σε ομοσπονδιακό επίπεδο στη Γερμανία για να βρεθεί μια λύση. Οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων για τον κανονισμό των ζωικών υποπροϊόντων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γερμανία και θα αναλαμβάνει δράση όποτε ε, υπο, στην προσοχή της ότι υπάρχει θέμα πλημελούς εφαρμογής των κανόνων. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υποθεί κάτι παραπάνω. Νομίζω οι αναφέροντε θα πρέπει να ψάξουν διαφορετικέ εναλλακτικέ λύσει να λύσουν το πρόβλημά του στο εσωτερικό τη Γερμανία. Ευχαριστώ πολύ. Θέλουν οι πολιτικές ομάδες να πάρουν το λόγο. Λίγα μπορούμε να πούμε, λέει η κυρία Μαέστρε, γιατί δεν έχουμε λάβει και πολλές πληροφορίες. Είναι πολύ δύσκολο να έχει κανείς θέση όταν δεν έχει λάβει κάποια έκθεση, έστω και μια τεχνική έκθεση που να μας επιτρέψει και μας να κρίνουμε με αρκετά στοιχεία ε, γιατί δεν ξέρουμε αν έχει λόγους και επιχειρήματα ο αναφερόμενος ή όχι. Πρέπει να μας στέλνετε τις πληροφορίες, γιατί δεν μπορούμε εμείς ως Επιτροπή να δράσουμε. Δηλαδή ούτε ως εκπρόσωποι της ΠΕΤΗ, ούτε ως βουλευτές, ούτε να μπορούμε να συντονίσουμε το τι θα γίνει με αυτές τις αναφορές, γιατί ακόμα δεν έχουμε λάβει καν την απάντηση από τις τοπικές αρχές. Σας ευχαριστώ πολύ. Η πρότασή μας είναι να μείνει ανοιχτή και να στείλουμε στις αρμόδιες εθνικές αρχές μια επιστολή για να μας απαντήσουν γιατί όπως είπατε κι εσείς δεν έχουμε απάντηση και χωρίς αυτήν δεν είμαστε σε θέση να αποφασίσουμε. Ούτε ξέρουμε αν πρέπει να κλείσουμε την αναφορά ή να την αφήσουμε ανοιχτή, να ζητήσουμε παραπάνω δράση. Λοιπόν, επιστολή προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές και παραμένει ανοιχτή. Περνάμε λοιπόν στο 13 που είναι 0248 του 19 από τον Μπενεντέτο Ρουμπέτη, Ιταλό υπήκο, ο οποίος είναι κατά της κατασκευής μονάδας αφαλάτωσης ε, για ανεξάρτητη παροχή νερού στο νησί της Έλμπα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο, ε, ο κύριος Καβαδάς από την Γενική Διευθυνσία μια και ο αναφέρον δεν βρίσκεται στην αίθουσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Και σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα να λάβω το λόγο. Ο αναφέρον εδώ εικάζει ότι η οικοδόμηση μονάδα αφαλάτωση στην Ίσο Έλβα στην Ιταλία θα δημιουργήσει περιβαλλοντικά προβλήματα. Έχουμε κοιτάξει το περιεχόμενο της αναφοράς και βάσει των όσων περιλαμβάνει ως περιεχόμενο, εξετάσαμε τις ε, διαδικασίες, την οδηγία για τα ύδατα, την οδηγία για την φύση και τις σχετικές όλες, τη σειρά οδηγιών και την περιβαλλοντική μελέτη αντικτύπου. Στην οδηγία για, την Natura, ε, για το Natura είδαμε το κατά πόσο είναι προστατευόμενη η περιοχή και ο τόπο που θα εγκατασταθεί η μονάδα θαλάτωση. Μετά για τα είδατα, ε, η εικασία ότι η μονάδα θα έχει αντίκτυπο στη μορφολογία της ακτής αλλά κοιτάζοντας τη, μορφή, τη μορφολογία των ακτών στην Ιταλία και βάσει των όσων προβλέπει ο οδηγία πλαίσιο για την προστασία των υδάτων, δεν βλέπουμε να προκύπτει εδώ θέμα. Εάν η μονάδα φαλάτωσης ε, οικοδομηθεί μακριά από την ακτή, ίσως να δημιουργηθεί πρόβλημα, διότι τα απόβλητα από την ε, επεξεργασία των υδάτων μπορεί να αποθέτονται στη θάλασσα αλλά υποθέτουμε ότι τα απόβλητα θα είναι αντικείμενο επεξεργασία κοντά στη μονάδα φαλάτωση, παρόλο που απέχει χιλιόμετρα από την ακτή. Παρόλο που αυτά τα στοιχεία δεν τα λαμβάνω τώρα αναφέροντα. Ε, οι μονάδε αφαλάτωση από τα παρατήματα 1 και 2 δεν καλύπτονται ε, από την παρεμβολική μελέτη αντικτύπου. Όμω τα κράτη-μέλη μπορούν να εφαρμόσουν αυστηρότερου κανόνε εφόσον το επιθυμούν για τη μελέτη αντικτύπου εντό μια δεδομένη χώρα, οπότε τίποτε δεν εμποδίζει τι Ιταλικές αρχές να ε, ολοκληρώσουν, να οργανώσουν μια περιβαλλοντική μελέτη αντικτύπου. Πάντως το συμπέρασμά μας είναι ότι βάσει των στοιχείων που έχουμε τώρα είναι ότι θα ήταν καλύτερο να φέρουν πρώτα απ' όλα να απευθυνθεί στις ε, Ιταλικές αρχές σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και να ε, συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό, για τη μονάδα φαλάτωσης. Θα έπρεπε να αναζητηθεί λύση σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Και αν αργότερα υπάρξει η σαφής εικόνα ότι βρίσκεται πρόβλημα, επανέλθει στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υποβάλει νέα αναφορά. Πολύ καλά. Κάποια πολιτική ομάδα Κύριος Κανίφ, ναι, ευχαριστώ πολύ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ε, εδώ δεν υπάρχει λόγος για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ίσως είναι η ευθύνη του αναφέροντα που δεν παρουσίασε κάποιες σχετικές πληροφορίες. Εδώ έχουμε τοπικές λεπτομέρειες πολύ συγκεκριμένες που παρουσιάζονται, τις οποίες εμείς δεν είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε Και νομίζω ότι δεν γίνεται να αξιολογηθούν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ θα προτείνω λοιπόν να κλείσει. Άλλος. Κυρία Μάιστρε. Δεν έχουμε την επιπτωσιολογική μελέτη, οπότε καλό θα ήταν να έχουμε αυτές τις πληροφορίες. Εγώ θα ήθελα να μείνει ανοιχτή μέχρι να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο. Εσείς θέλετε να κλείσει. Όχι. Δεν το είπα καλά. Αυτό που λέω είναι αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά περισσότερες πληροφορίες από τον αναφέροντα, ε, μέχρι να στείλει όλα τα σχετικά στοιχεία, για να δούμε μήπως έχει αυτή η μονάδα φαλάτους αρνητικές συνέπειες για την περιοχή, να ζητήσουμε να μας στείλει και εμάς πληροφορίες, να τις μελετήσουμε και μετά να αποφασίσουμε αν θα κλείσουμε. Αλλά πριν κλείσουμε, να δώσουμε τη δυνατότητα να στείλουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά. Ωραία. Λοιπόν, την αφήνουμε ανοιχτή, αλλά με προθεσμία μια και ο αναφέρον δεν απάντησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε, εφόσον ενεργοποίησε την αναφορά, απαιτούμε από τον ίδιο να μας στείλει νέα στοιχεία μέσα σε δύο μήνες από τη στιγμή που θα λάβει την επιστολή μας και μετά θα το κλείσουμε μέσα σε μια συνάντηση συντονιστών. Και μετά έχουμε τη τελευταία που είναι στην ημερήσια διάταξη. Η Μανουέλα Τζακομίνη από το Animal Welfare ε, ε, Foundation για τα, ε, τις εκμεταλλεύσεις αίματος και για τις εγγύους φοράδες και τον ορό γονοδοτροπίνης. Έχετε πέντε λεπτά. Και μετά, αφού σας ακούσουμε, και ακούσουμε και τις πολιτικές ομάδες. Ε, θα σας δώσουμε άλλα δύο λεπτά ε, για τα συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ. Κυρία Γκούρτνερ, νομίζω. Ναι, ωραία. Έχετε το λόγο. Thank Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την δυνατότητα να μιλήσω σήμερα. Εργάζομαι για οργάνωση για την προστασία των ζώων στην ε, Αργεντινή και τον Ουρουάη από το 2015. Πρέπει να ξέρετε ότι παίρνουμε ορό από το αίμα των φοράδων για να δημιουργηθεί το PMSG που χρησιμοποιείται σε φάρμακα και την ιατρικά. Δεν βλέπω να λειτουργεί το σύστημα με το τηλεκοντρόλ που έχω εδώ. Δεν βλέπω να μπορώ να προχωρήσω τις διαφάνειες. Χρειάζομαι βοήθεια παρακαλώ. Μία από τις μεγαλύτερες ε, ανησυχίες μας είναι η κακομεταχείριση των φοράδων και επίσης ο μεγάλος όγκος και η συχνή λήψη αίματος από τις φοράδες. Μέχρι 10 λίτρα κάθε εβδομάδα αφαιρούνται. Μετά από 4 μήνες εγκυμοσύνης, όταν το επίπεδο του PMSG πέφτει, τότε δημιουργείται τεχνητά άμβλωση στις φοράδες για να μπορέσουν να ξαναμείνουν σε κατάσταση εγκυμοσύνης. και χωρίς μάλιστα την κατάλληλη επίβλεψη πάντα. Δεν καταφέρνω να προχωρήσω τις διαφάνειες όπως πρέπει. Τρίτη διαφάνεια. Μπορείτε να με βοηθήσετε να πάμε στην τρίτη διαφάνεια. Α, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, οι έρευνές μας από το 2018 δείχνουν ότι η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί τα τελευταία τρία χρόνια. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι δεν είναι δυνατόν, δεν είναι εφικτό να υπάρξει μεγάλη ε, σημαντική βελτίωση. Εξάλλου αυτά τα αγροκτήματα του αίματος είναι πολλά και είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκπαιδεύσουμε κατάλληλα αυτούς που χειρίζονται τις φοράδες ώστε να μπορούν να τις χειρίζονται χωρίς να δημιουργούν πόνο. Έπειτα είναι το θέμα της εγκαιμοσύνης που είναι δύο φορές το χρόνο και είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιβλέψει κανείς τι γίνεται με τις φοράδες γιατί κρατούνται συνήθως σε μέρη μέσα στα δάση ή σε ακροκτήματα που είναι δύσκολο να έχει κανείς πρόσβαση. The import of PMSG from South America should... Πρέπει να σταματήσει η εισαγωγή λοιπόν του PMSG από την Νότια Αμερική. Δεδομένη τη της κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι φοράδε, ότι δεν υπάρχει κτηνιατρική επίβλεψη επίσης ούτε τα αγροκτήματα αυτά ε, επιβλέπονται από τις αρχές. Επίσης δεν τηρούνται οι συμφωνίες που λένε ότι τα συμβαλόμενα μέρη μπορούν να υιοθετήσουν μέτρα για να προστατεύσουν ε, τη δημόσια ηθική και να προστατεύσουν και την προστασία των ζώων ή την υγεία των ζώων. Θέλω λοιπόν να τονίσω ότι το 2009 η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε την εισαγωγή προϊόντων από για λόγω προστασίας των ζών. Θέλω λοιπόν να ζητήσω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προωθήσει την απαγόρευση της εισαγωγής του ορού αυτού από τη Νότια Αμερική, δεδομένου ότι κάπου 2 εκατομμύρια πολίτες έχουν υπογράψει σε συγκέντρωση υπογραφών για να μην ε, γίνεται αυτή η εισαγωγή. Εξάλλου παραβιάζεται η ευρωπαϊκή, νομοθεσία και υπάρχουν ήδη συνθετικά προϊόντα που μπορούν να αντικαταστήσουν την ε, γόνατα τροπίνη του ορού εγγύου φοράδας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ε, αναφέρουσα. Πολιτικές ομάδες τώρα θέλουν να πάρουν το λόγο. Α, όχι, πρώτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγγνώμη. Πρώτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ο κύριος Στάνης Λαφράτσε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και καλησπέρα περίπου. Καλό βράδυ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει ότι πιθανόν οι φοράδες ε, να μην τυχαίνουν καλή συμπεριφορά εξαιτία της γοναδοτροπίνης ε, του ορού τους και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάποιους συνομιλητές και έχει έρθει σε επαφή και με ε, τους αναφέροντες. Θέλω πάντως να σας υπενθυμίσω ότι οποιασδήποτε προδιαγραφές επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των ζώων που επιβάλλει αλλού πρέπει να συνάδουν και με τους κανόνες του ΠΟΕ. Όμως οι διεθνείς ε, ανταλλαγές που γίνονται λαμβάνουν υπόψη ε, τα μέτρα τα υφωτογειονομικά που περιλαμβάνονται στους κανονισμούς του ΠΟΕ. Τώρα για την παραβίαση της νομοθεσίας εδώ θέλω να πω ότι η νομοθεσία για την προστασία των ζώων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζεται μόνο στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια και δεν είναι δυνατόν να επιβάλλουμε τέτοιες ε, συνθήκες αλλού για τέτοια προϊόντα ή για παράγωγά τους. Αυτό πρέπει να είναι σαφές. Εξάλλου η Ευρωπαϊκή του. δεν μπορεί να ειναι σαφε εξαλλου η ευρωπαικη ενωση δεν μπορει να επιβαλλει σε τρίτε χώρε τι προδιαγραφέ τη και πρέπει να σέβεται και του κανονισμού του ΠΟΕ. Και παρόλο που η Επιτροπή δεν προτίθεται να απαγορεύσει αγωγέ γονοδατροπίνε του ορού εγγύου πιστεύει ότι οι χώρες της Νοτιοαμερική θα πρέπει να εξασφαλίσουν ικανοποιητικό επίπεδο εφαρμογή των διεθνώ συμφωνημένων αρχών και προτύπων για την καλή διαβίωση των ζώων του ΠΟΕ. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται ώστε να βελτιωθούν οι προδιαγραφές αυτές. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, οι βουλευτές παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τους αναφερόμενους. και όλους στην Ευρώπη που υπέγραψαν αυτή την αναφορά. Είναι δύσκολο να μην επηρεάζεται κανείς ε, παρακολουθώντας αυτό το βίντεο για το πώς ε, αντιμετωπίζουν ε, τα άλογα στην Αργεντινή και στην Ουρουγουάη. Η ερώτησή μου είναι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόσφατα έκλεισε η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ για εμπορικά θέματα και αυτή η συμφωνία προφανώς έχει ε, και τα ε, κεφάλαια σχετικά με τα υγειονομικά και φυτογειονομικά ε, θέματα. Φαντάζομαι πως ο ευρωπαϊκός πληθυσμός ανησυχεί αρκετά όταν στα πλαίσια των βαθύτερων εμπορικών σχέσεων δεν χρησιμοποιείται το πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωση Μερκοσούρ για να αντιμετωπίσουμε θέματα ευζοία των ζώων, τουλάχιστον ε, στα θέματα που είναι στο κεφάλαιο για τα υγειονομικά και ε, φυτοϊγειονομικά θέματα. Έχουμε σχέσεις με τις χώρες αυτές και στα πλαίσια αυτών των σχέσεων θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε αν έχει τεθεί το θέμα στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων στη συμφωνία με τη Μερκοσούρ και αν όχι για ποιο λόγο δεν ετέθη. Πιστεύω πως ως Επιτροπή Αναφορών καλό είναι να στείλουμε ε, αυτή την ε, αναφορά στην Ίντα, την Επιτροπή Εμπορίου και να δούμε αν ε, μπορεί να το δει υπό το φως των διαπραγματεύσεων που τρέχουν και των σχέσεων που έχουμε των εμπορικών με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής για να δούμε ενδεχομένως τι δράση θα μπορούσε να αναλάβει για το θέμα αυτό, για την απαγόρευση εισαγωγών για παράδειγμα για τα προϊόντα που προέρχονται από φώκες. Ε, χρειάστηκε να περάσουν πάρα πολλά χρόνια, πολύ πολιτική πίεση ασκήθηκε, δεν γίνονται αυτά από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά επειδή ακριβώς ε, θα ε, εμβαθυνθούν ενδεχομένως τα εμπορικέ μα σχέσει με τι χώρε αυτέ, ίσω θα έπρεπε το θέμα να το δούμε από αυτή την οπτική γωνία. Πριν δώσουμε το λόγο σε άλλους ευρωβουλευτές, να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, απαντήσει στην κυρία Ντάρλινγκ για το κατά πόσο η συμφωνία με τη Μερκοσούρ έχει ε, συμπεριλάβει και τέτοια θέματα. Θεωρώ πως είναι πολύ λογικό και συμφωνώ με τη συνάδελφο. Ωραία λοιπόν, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ που μου δώσατε και πάλι το λόγο και ευχαριστώ για την ερώτηση για τις διαπραγματεύσεις αυτές εμπορικές. Θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τη Γενική Διεύθυνση Trade Εμπορίου Δράτω με τις ευκαιρίες για να σας υπενθυμίσω πως για τα πρότυπα και τους κανόνες για την ε, ευημερία των ζώων δεν έχουμε δικαίωμα να επιβάλλουμε ε, προϋποθέσεις κατά τις εισαγωγές, αλλά οι διαπραγματεύσεις είναι αμφίδρομες, οπότε θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να συμφωνήσουν και να ενισχύσουν τα πρότυπα αυτά στα πλαίσια της συμφωνίας μας. Αυτό έχω να πω, όχι κάτι άλλο. Κυρία Εύη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ ήθελα το λόγο για να εκφράσω θερμές ευχαριστίες προς τους αναφέροντες. Φύγουν ένα θέμα που πραγματικά είναι φρικτό. Δεν μπορώ να το πω αλλιώ. Είναι φρικτό. Ακούσαμε ότι δεκάδες χιλιάδες έγκυοι φοράδες αναγκάζονται να υποβληθούν σε λήψη αίματος για να παραχθεί αυτός ο ορός, ο στην Ευρώπη. Η βαρβαρότητα αυτή γίνεται πραγματικά πραγματικότητα στα αγροκτήματα αίματος, όπου οι φοράδες υποβάλλονται σε επανειλημμένες εγκυμοσύνες και αμβλώσεις θα μπορούσαν να αναζητηθούν συνθετικές, χημικές εναλλακτικέ για να μην υποβάλλονται τα ζώα σε, αυτές, σε αυτά τα περιτά βασανιστήρια. Είναι όμως ε, αμήλικτα και ανελαίητα τα συμφέροντα των φαρμακευτικών εταιριών. Ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει από καιρό ότι επειδή όλα αυτά συμβαίνουν από την άλλη πλευρά του ωκεανού, δεν υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν. Εμείς όμως γνωρίζουμε ότι αυτό δεν αληθεύει. Εργαλεία υπάρχουν. Εάν όμως έχουν δικαίωμα εξαγωγών αυτέ οι μονάδε προ την Ευρωπαϊκή Ένωση από του ίδιου του φορεί που αποτίθεται ότι του παρακολουθούν. Δεν υπάρχει κανένα έλεγχο. Αυτά τα αγροκτήματα αίματο και κτηνίατροι δεν έχουν την παραμικρή δυσκολία στην εξάσκηση των δραστηριοτήτων του. Δεν είναι δυνατόν να ε, βασανίζεται νομίμω ε, μια φοράδα σε όλη τη διάρκεια τη ζωή τη για να αυξάνεται τεχνητό η γονιμότητά τη και να υπάρχουν απεριλημμένες εγκυμοσύνε πριν οδηγηθεί στο σφαγείο είναι ένα ε, στρεβλό και ανώμαλο μοντέλο κτηνοτροφία, το οποίο θα οδηγούσε σε αγανάκτηση όλου του Ευρωπαίου πολίτε, αν το γνώριζαν. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρξει απαγόρευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτών των προϊόντων με το συγκεκριμένο ορό τη γοναδοτροπίνη από την Νότια Αμερική. Το έχω πει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ρώτησα και τον περασμένο μήνα, αλλά διαρκώ αποντά όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα έλεγα λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει να προχωρήσει αναφορά αυτή και να ζητήσει απαγόρευση αυτή τη ουσία στην Ευρώπη. Είναι η μόνη νόμιμη οδό που θα μπορούσε να συμβάλλει στο να δοθεί ένα τέρμα σε αυτό το βασανιστήριο που, οδηγεί, που προκαλεί τόση, ε, τόσο πόνο αυτό το αιματοκύλισμα των ζώων. Ε, θα συμφωνήσω λοιπόν με όσα είπε και η συνάδελφος Κίλτον Ντάρλι. Καλό είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΙΝΤΑ να λάβει γνώση του συγκεκριμένου θέματος και να κοιτάξει να ε, μελετήσει περαιτέρω και να φωτίσει τις εμπορικές μας σχέσεις με την Νότια Αμερική ακόμη και στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Μερκοσούρ θα έλεγα συντονιστές της Επιτροπής μας να προτείνουν προφορική ερώτηση ή έστω ένα ψήφισμα από του θέματος, ώστε το Κοινοβούλιο να πάρει σαφή θέση υπέρ μιας απαγόρευσης αυτών των προϊόντων στην Ευρώπη. Υπάρχει δυνατότητα να το κάνουμε. Οπότε νομίζω ότι ηθικώς ε, έχουμε την επιταγή να το κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Εσείς όχι. Ωραία λοιπόν. Για να κλείσουμε το θέμα θα το λόγο στην αναφέρουσα για δύο λεπτά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ευρωβουλευτές που στηρίζουν την αναφορά. Είμαστε σε συνεχή επιτροπή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό, από το 16 και μετά, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά πάντα, αλλά με τρόπο που είναι ατελής ή μη ικανοποιητικός. Για παράδειγμα, προτείναμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσουν από την ΕΦΣΑ να γνωμοδοτήσει για τα θέματα αυτά παραγωγής του της ορμόνης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε αυτό είναι εκτός αρμοδιότητας της ΕΦΣΑΣ. Παρ' όλα αυτά έχει σχετικές ε, διατάξεις ε, για την ευζοία των ζών ε, ζώων και έχει τη δυνατότητα να γνωμοδοτήσει για θέματα ασθενειών και ευζοίας. Το 2017, για παράδειγμα, γνωμοδότησε γραπτά για το κυνήγι της φώκιας και η επιστημονική αυτή έκθεση μαζί με τις ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών ήταν ουσιαστικέ στη μακρά διαδικασία που οδήγησε στην απαγόρευση εισαγωγή τέτοιων προϊόντων ε, του 9. Άρα λοιπόν ο Καναδάς κατέθεσε ε, αγωγή στον ΠΟΕ ε, εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, η Σχετική Επιτροπή του ΠΟΕ στήριξε την απαγόρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπε πως είναι απαραίτητη για να στηρίξει τη δημόσια ηθική σε θέματα προστασίας ε, της ευημερίας των ζώων. Επίσης, η χρήση των ζώων στην παιδεία και στην έρευνα. Αυτό θα έπρεπε να καλύπτει και τις φοράδες αυτές ε, όμως οι διατάξεις δεν έχουν ε, τέτοιου είδους αρμοδιότητα γιατί το αίμα αυτό δεν, δεν ε, αφαιρείται για επιστημονικούς λόγους αλλά για οικονομικούς, ξεκάθαρα. Το 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι θα έπρεπε από αυτά τα αγροκτήματα παραγωγής αίματος ε, να ε, συμπεριληφθούν σε ελέγχους που γίνονται στην Αργεντινή και στην Ουρουάη αλλά ακόμα αυτό δεν έχει γίνει. Επίσης Υπάρχει μια εταιρεία στην Ουρογουάη που τη λένε Syntax που εξάγει τέτοιου είδους ε, ορμόνες στη Γαλλία παρόλο που δεν είναι εγκεκριμένος φορέας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε ε, ενημερώσει και τις γαλλικές αρχές και την ευρωπαϊκή αλλά αυτή η παράνομη εισαγωγή του της ορμόνης συνεχίζεται. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Πρώτα απ' όλα, η πρότασή μας είναι να αφήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά. Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει σε επαφή με τη Γενική Διεύθυνση Trade, να δει τι γίνεται στα πλαίσια της Εμπορική συμφωνίας με τη Mercosur, να δούμε μέχρι πού έχουν φτάσει οι διαπραγματεύσεις για τα θέματα αυτά, τα υγειονομικά, τα φυτογειονομικά, προστασία των ζώων και θα ζητήσουμε από την Επιτροπή Ίντα που παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας με τη Μερκοσούρ για να μας στείλει πληροφορίες σχετικά και τρίτον Επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει πως η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάντα θα σέβεται τις διατάξεις του ΠΟΕ, και οι έλεγχοι θα γίνονται στην τρίτη χώρα και επίσης πως οι διατάξεις για την προστασία των ζών θα πρέπει ε, να προστατεύονται από την αντίστοιχη ε, Διεθνή Επιτροπή. Θα ήθελα να έχουμε μια γνωμοδότηση της Επιτροπής αυτής και του ΠΟΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει αρκετές συναντήσεις με τις αρχές των χωρών αυτών, των χωρών ε, προέλευσης Στην απάντησή τη σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα είπε πολλές φορές πως θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία οι χώρες προέλευσης, όπως επίση και με τους κανόνες τη Διεθνού Επιτροπής και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Θα του ζητήσουμε λοιπόν να μας πούν τι γίνεται. ενημερώνοντά του πώ έχουμε αρκετέ αναφορές, ε, αρκετού αναφερόμενου που ζητούν να λύσουμε το θέμα. Για το λόγο αυτό λοιπόν θα ζητούσαμε τα συγκεκριμένα που σας προανέφερα. Θα αφήσουμε την αναφορά ανοιχτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν δεν κάνω λάθος, τελειώσαμε. Κυρία Εύη. Μόνο το εξή να προσθέσω. Αν γίνεται να το στείλουμε και στην διακομματική ομάδα για τα ζώα. Την έκθεση αυτή. Την αναφορά αυτή. Ναι, ναι, βεβαίως. Οπότε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι λίγη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών. Συνεχίζουμε αύριο το πρωί με τους συντονιστές. και με τους αναφέροντες.